Θα ήθελα να σας μιλήσω ότι μιλούμε τώρα για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021 με 2027. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι το σχέδιο γνωμοδότησης ε, το εξετάσαμε το Σεπτέμβριο στην ε, ομάδα μας στην Επιτροπή μας και είχαμε 247 ε, τροπολογίες. Έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας για αυτό το θέμα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Μλίναρ, για 5 λεπτά. Παρακαλώ πολύ να τηρήσετε το χρόνο σας, γιατί έχουμε πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα παραμείνω στα 5 λεπτά και νομίζω ότι και τα 40 λεπτά θα μας φτάσουν για να συζητήσουμε το πρόβλημα. Λοιπόν, το θέμα αυτό. Να σας πω καταρχά με καθαρή συνείδηση και με μεγάλη ικανοποίηση ότι το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη έχει δημιουργήσει μια πολύ θετική συζήτηση με τους κοιόδης εισηγητές και ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στην, ε, στην ε, ε, σύνταξη των τροπολογιών. Στις 26 Σεπτεμβρίου είχαμε την πρώτη συνάντηση σκιωδών. Ορίσαμε μία εντολή για να συζητήσουμε σε επόμενες τεχνικές συναντήσεις. Δύο, μία αύριο και μία την επόμενη εβδομάδα. Να τονίσω ε, εν συντομία ότι ένα βασικό στοιχείο της πρότασης δεν αμφισβητήθηκε στο σχέδιο έκθεσης ούτε από τις ε, τροπολογίες ε, τις πολλές τις οποίες ε, κατέθεσαν οι πολιτικές ομάδες ε, που είναι ο συνολικός προπολογισμό για το πρόγραμμα. Όπως ε, προέκυψε κατά την προηγούμενη συζήτηση, το 9,2 δις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να θεωρηθεί κατά τις ε, προσεχείς διαπραγματεύσεις ως ελάχιστο ποσό που θα μας εξασφαλίσει την επιτυχή έκβαση του προγράμματος και εφαρμογή του. Ένα ακόμη βασικό ζήτημα είναι ο συνολικός στόχος του προγράμματος και ε, ο καθορισμός του πεδίου εμβέλειάς του και της επιλεξιμότητας για συμμετοχή. Εστίασε συγκεκριμένα στην προστιθέμενη αξία του προγράμματος και την ευαισθησία τομέων όπως ε, κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη θα λάβουμε υπόψη ε, όλες τις συνεισφορές ε, για να υπάρξει μια εξισορροπημένη ε, λύση για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες απλοποίησης και ευελιξίας όσον αφορά την τεχνογνωσία και την πρόσληψη αυτής ώστε τα προγράμματα που θα χρηματοδοτήσει αυτό το πρόγραμμα να μην απειλήσουν ε, την ε, ασφάλεια της Ευρώπης. Ε, η τεχνητή νοημοσύνη επίσης είναι σημείο που θα προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως. Οι τροπολογίε από όλε τι πολιτικές ομάδες αναφέρθηκαν στους κόμβους ε, καινοτομία, που ήταν πολύ σημαντικό ζήτημα από, τη δημοσίευση της πρότασης και εξή. Θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καθαρότερη εικόνα, ώστε να υπάρχει, ώστε η δημιουργία του ε, δικτύου κόμβων να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Η μία πτυχή θα εξασφαλίζει την εφαρμογή τη ανάπτυξη. Ε, του προγράμματος ε, με ευελιξία ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ αυτού του προγράμματος και άλλων πηγών χρηματοδότησης. Δεύτερον, οικοδόμηση επί της ε, υφιστάμενης υποδομής και προηγούμενων αναλογικών, μάλλον ανάλογων ε, εμπειριών όπως το πρόγραμμα Horizon 2020, διάβλη συνεργασία μεταξύ ε, των κόμβων καινοτομία και του προγράμματο Ψηφιακή Ευρώπη αλλά και άλλων φορέων. Επίση, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο στόχος του προγράμματο αυτού και ε, των πόρων του δεν θα χαθεί και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χάσει μία καλή χρονική στιγμή και την κεκτημένη ταχύτητα που υπάρχει ε, για την ψηφιοποίηση. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η συζήτηση στις ε, επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν. Μέχρι τώρα ήταν πολύ καλή συνεργασία και μέχρι τότε ήταν πολύ καλή συνεργασία και οι άλλες επιτροπές ε, τήρησαν το χρονοδιάγραμμα και εκείνες. Πρόεδρος, μπράβο σας. Είστε ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα φυσικής νοημοσύνης. Η κυρία Δελκαστήγιο. Έφτασα. Τα κατάφερα. Συζητήσαμε ε, με την συνάδελφο ε, περπατώντας, οπότε δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, δεν χρειάζεται να το πω, ούτως ή άλλως το έχουμε πει αυτό. Ως, ε, όπως ε, είπε και η συγγήτρια, θα ήθελα να, να υποστηρίξω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όταν θα υπάρξει η ανάγκη αύξηση των προτεραιοτήτων πέρα από την κυβερνοασφάλεια και τις σχετικές υποδομές. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην υπάρχει ένα ευχολόγιο ατελείωτο για να μην χαθούν τα κονδύλια που θα κάνουν την πραγματική διαφορά. Θα ήθελα δύο πτυχές να αναφέρω που η συγκήτρια γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έχω μάλιστα υποβάλει και σχετική τροπολογία. Το ένα είναι όσον αφορά την επέκταση του προγράμματος ικανοτήτων σε τρίτη χώρα. Ο, ε, ε, πρέπει να αρχίσει η συζήτηση. Νομίζω όμως ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια εξισορροπημένη προσέγγιση ώστε το επίπεδο συμμετοχής των τρίτων χωρών ε, να εξετάζεται κατά περίπτωση βάσει των στόχων, σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού. Και τέλος, όσον αφορά τη διοντολογία και την τεχνητή νομοσύνη εγώ υποστηρίζω το πρόγραμμα, όμως πρέπει κάπως να το επεξεργαστούμε, να το τελειοποιήσουμε γιατί η ιδεοντολογία αφορά σε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο πρόγραμμα Horizon. Ε, πρέπει να πω ότι η συνεργασία με την εισηγήτρια ε, πηγαίνει πολύ καλά. Είμαι μία από τις ε, σκιώδεις ε, ε, εισηγήτριες. Κάποια πράγματα πρέπει να τα προσαρμόσουμε, να τα αναδιατυπώσουμε, αλλά νομίζω ότι πραγματικά θα είναι πάρα πολύ εξαιρετική η έκβαση με τη δουλειά της εισηγήτριας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντελκαστήγιο και τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Ζωρίνιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν σχέσεις και δεσμοί στην ψηφιακή τεχνολογία και στις διάφορες χώρες. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα για ψηφιακή Ευρώπη. Έχουμε κοινέ αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση αυτές πρέπει να μπούμε στην μπροστοφυλακή του ψηφιακού κόσμου. Υπάρχουν πολλές προτεραιότητες, αλλά είναι λίγο ασαφής πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι εις ό,τι αφορά την οργάνωση της ε, διασφαλίσης του προϋπολογισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι πολύ φιλόδοξο και με βάση το χρονικό ορίζοντα. Είναι εξαιρετική η συμβολή της εισηγήτριας σε όλα αυτά τα θέματα και τη συγχαίρω. και άλλοι εισηγητέ συνέβαλαν ώστε να έχουμε ένα στιβαρό μέσο για πρόοδο. Ε, έχουμε καταρχήν το θέμα της συνεργασίας ώστε να υπάρχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες στον ψηφιακό κόσμο χωρίς απώλεια ελέγχου περιεχομένου. Πρέπει να δούμε τις επιδόσεις και την ασφάλεια στον κυβερνό χώρο και το άλλο θέμα είναι πώς θα, ε, δια, ε, θα κάνουμε ε, διαφανές το πρόγραμμα σε σχέση και με άλλα χρηματοδοτικά, να προλάβουμε συστημικές εκπτώσεις, ε, επικαλύψεις και τέλος ε, ποιο θα είναι το ηθικό περιεχόμενο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε και το ηθικό, δεοντολογικό περιεχόμενο της ψηφιακής μετάβασης στην Ευρώπη. Πρέπει να προσπίσουμε τις αξίες της Ευρώπης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ασφάλεια, ε, προστασία, πρόσβαση, καθολικότητα. Ε, περίπου 300 τροπολογίες υπευλήθησαν. Πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά χρειάζεται να βρεθεί μια ισορροπία στο κείμενο και να προσέξουμε τα βασικά θέματα. διασφάλισης, συνεργασίας δηλαδή με τρίτες χώρες, με βάση τα ορθά κριτήρια και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και να ε, ολοκληρώσουμε την ανάπτυξη ε, στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Άσλι Φόξ για τους Ευρωπαίους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές στο ΙΤΡΙΤΗ σε μέγεθος ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, γεγονός είναι αυτό. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την συνεργασία της στο φάκελο αυτό. Το πρόγραμμα ψηφιακής Ευρώπης είναι πολύτιμη πρόταση που θα βοηθήσει οι επιχειρήσεις, τη δημόσια διοίκηση, να ε, προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο, στην οικονομία και την κοινωνία, νέες ειδικότητε για νέες θέσεις εργασίας, για να δράξουν τις ευκαιρίες της νέας οικονομίας ε, που θα γίνει έτσι πιο δυναμική και ανθεκτική. Οι επιχειρήσεις θα λύσουν θέματα κυβερνοασφάλειας, θα αναπτύξουν νέες αγορές, θα αυξήσουν τις εξαγωγές, θα βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση, θα γίνει πιο υπόλογη, αποτελεσματική μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα αναβαθμίσουν την ποιότητα για τους πολίτες. Ε, έχουμε ε, κέντρα ε, ψηφιακά. Ε, τα καλωσορίζομαι. Επίσης ε, καλωσορίζομαι την πρόσβαση στα δεδομένα. Η βελτίωση του συντονισμού με άλλα δίκτυα είναι σημαντική. Τώρα υπάρχουν κάποιες ασάφειες στην υλοποίηση. Για παράδειγμα, τα προγράμματα ανάθεσης ε, πρέπει να διευκρινιστούν. Ε, μας αρέσουν νέες προτάσεις για το στόχο της κυβερνοασφάλειας, αλλά βέβαια πρέπει να δούμε και τις προτάσεις της Κομισιόν που δεν τις είδαμε ακόμη. Ε, ο ρόλος μας δεν είναι σημαντικός. Η εισηγήτρια θέλει άμεση διαχείριση ε, για την για τη διαλειτουργικότητα και την εφαρμογή των ψηφιακών ειδικοτήτων. Τέλος, η πρόταση, κατά τη γνώμη μας, ε, ε, έχει στόχο βιομηχανικό και όχι στρατηγικό. Πώς οι τρίτες χώρες και οι ενώσεις τους ε, με βάση ισόρροπης συνεισφοράς θα βελτιώσουν τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Επίσης, πολέμηση του προστατευτισμού. Η κοινή, το κοινό εγχείρημα για υψηλή ταχύτητα, υπολογιστές είναι το βασικό μέσον για την αναβάθμιση των υπολογιστών και έτσι θα ανοίξουν οι ορίζοντες. Αν όμως μια τρίτη χώρα είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο αυτό αλλά όχι με την ψηφιακή Ευρώπη, η... Γενικά συμφωνεί η ομάδα μου με την πρόταση κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε την εισηγήτρια για τις προσπαθειές της. Ευχαριστώ Ashley. Ε, δεν βλέπω να υπάρχουν όλοι. Πάμε στον κύριο Μπιουτικόφερ από τους Πρασίνους. Που είναι όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, την πέμπτη μεγαλύτερη ομάδα και στο Κοινοβούλιο και η περήφανη που ε, είναι στην, ε, στο Κοινοβούλιο έτσι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια καθώς επίσης και τους σκιώδης ε, για αυτήν την πολύ παραγωγική και επικοδομητική συνεργασία. Εγώ θα ασχοληθώ με μικρότερα ας πούμε, σημεία τα οποία ακόμα ε, βρίσκονται υπό συζήτηση και υπό διαπραγμάτευση. Πιστεύουμε ότι η ηθική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης ε, είναι πολύ σημαντική και ε, ακούμε ότι θα προσθεθεί μια μικρή παράγραφος εδώ και είναι πολύ καλό. Επίσης, βλέπουμε μια ψηφιακή απόκληση όχι όμως μόνο μεταξύ των διαφόρων χωρών αλλά και μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό αυτή η δεύτερη απόκληση, αυτό το δεύτερο κενό ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεπεραστεί. Ε, η ψηφιακή καινοτομία ε, βοηθάει, πρέπει να παίξουμε σημαντικό ρόλο και στο σημείο αυτό και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτά τα hubs στην ουσία είναι οικοδομημένα με παρόμοιο τρόπο και ε, με παρόμοια πρότυπα στις διάφορες περιφέρειες και στις διάφορες χώρες. Δηλαδή παντού να είναι ίδιο το σκεπτικό τους. Έχω κάποιο προβληματισμό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν προσπαθεί να περιορίσει το πρόγραμμα ε, ε, ψηφιακής Ευρώπης ε, ξέχωρα και πέρα από το Κοινοβούλιο. Αυτό δεν είναι καλή εταιρική σχέση με το Κοινοβούλιο. Τέλος, το ζήτημα του ποιος θα έχει δυνατότητα συνεργασία συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Κατά την άποψή μου, κύριε Φόξ, αυτό το σημείο έχει στρατηγική σημασία. Και, κοιτώντας λίγο πιο πίσω, ας πούμε μια εβδομάδα πριν ε, ε, τη, τα θέματα κυβερνοασφάλειας ε, τα οποία ανακοίνησε το Bloomberg ε, που έδειξε ότι η τεχνολογία θα έχει δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, θα του δώσει λέω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει προωθημένη τεχνολογία, ούτως ώστε να ελέγξει εγκαταστάσεις ε, τεχνολογικές, βιομηχανικού ή άλλου τύπου, από μακριά, μέσα από το cloud και τα Επομένως η κυβερνοασφάλεια κατά τη δική μου άποψη είναι πυρηνικό σημείο και πυρηνική ανάγκη και επομένως θα πρέπει όσο περισσότερο και όσο καλύτερα μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό. Ε, ναι, μπορούμε να διευρύνουμε, αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν θα επιτρέψουμε οποιαδήποτε αποτυχία ε, ή παρίσφρηση όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπουτικόφερ γιατί ξεπεράσατε περίπου 63% τον χρόνο που σας είχαμε δώσει. Το λόγο... Το... Ε... only the fifth largest group, I may, may this. Σας έδωσα όμως ε, ε, λίγο χρόνο παραπάνω. Ε, μπορώ να μιλήσω και εξ της τη ΓΚΟΕ, δηλαδή να πάρω το χρόνο και τη ΓΚΟΕ. Ναι, δεν βλέπω κάποιον από την ΓΚΟΕ, αλλά από το FTD ο κύριο Σταμπουράνο. Εγώ όμω είμαι από πολύ μικρή ομάδα, δεν πειράζει. Είμαστε ικανοποιημένοι από με την εργασία τη συγγετρίας, την οποία ευχαριστούμε για το πνεύμα στην εργασία. Στο πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη είναι ένα θέμα που μα παθιάζει και μα συγκινεί. Ωστόσο υπάρχουν κάποια στοιχεία προβληματικά, τα οποία θα πρέπει να εμβαθυνθούν και να αντιμετωπιστούν. Ε, κατά την έννοια αυτή έχουν υπεβάλει τροπολογίε. Οπωσδήποτε υποστηρίζουμε το ψηφιακό πρόβλημα, αυτό είναι ένα αμφίβολο, θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ε, πολίτες ε, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και στο ύψος του διεθνούς ανταγωνισμού. Βεβαίως θα θέλαμε περισσότερη διαφάνεια ε, μεγαλύτερη συνέχεια στη δράση και μεγαλύτερη συμπερίληψη ε, και βεβαίως ε, προστασία της και σημασία στην γεωγραφική ισορροπία. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να μειωθεί αυτό το κενό το οποίο υπάρχει. Από την άλλη πλευρά το θέμα της κυβερνοασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η χρηματοδότηση των υποδομών που θα σώσουν δώσουν ε, ζωές και δεδομένα που θα είναι τα στρατηγικά μας asset πρέπει οι Ευρωπαίοι να αποκτήσουν ε, και να οικοδομήσουν ευρωπαϊκές ικανότητες. Άρα θα πρέπει ε, τα δημόσια κονδύλια τα οποία αφορούν την κατάρτιση, την ε, ανάπτυξη δεξιοτήτων να αυξηθούν έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ικανός πληθυσμός αρκετά προετοιμασμένος. Κατά την έννοια αυτή εμείς έχουμε άλλον ένα ισχυρό προβληματισμό όσον αφορά την digital addiction ε, την προσκόλληση δηλαδή αυτή ε, προς τον εθισμό στα ψηφιακά ε, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να το αποφύγουμε και άρα το πρόγραμμα να χρησιμοποιήσει αυτές τις ικανότητες. Εμείς έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και να προστατήψουμε τον κυβερνοχώρο και τους πολίτες μας. Τέλος, η εξέταση της λεγόμενης τεχνοηθικής, ε, τεχνολογικής της τεχνολογίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, για μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όλο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Γκρίφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάντα όταν ε, ε, υπάρχουν εκπρόσωποι της δεύτερης μεγαλύτερης ε, ομάδας. Εν περιπτώσει το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και στα πλαίσια του ορίζοντα Ευρώπη έχουμε πει ότι πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί και βεβαίως η συνάδελφος έκανε όπως πάντα μια πάρα πολύ καλά, καλή και ε, λεπτομερή δουλειά. Αλλά όπως είπε και ο Ντάριο προηγουμένως, ε, η ψηφιακή τεχνολογία είναι ένας τρόπος να προωθήσουμε και πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν μένει κανένας πίσω λόγω της ηλικία του, λόγω του ότι μένει ενδεχομένως στην Ήπεθρο ή σε ένα πιο απομονωμένο ε, μέρος. Θα πρέπει να καταρτήσουμε και να επανακαταρτήσουμε ε, όλο το εργασιακό δυναμικό η ψηφιακή ε, οικονομία καθώς επίσης ε, και οι καθαρές μορφές ενέργειας είναι μέρος ενός συνόλου. Ε, είναι αυτό που αφορά τον κόσμο, τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρίφιν. Άλλος κανείς ζητεί το λόγο. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Παντίκ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Κομισιόν ευχαριστώ την εισηγήτρια για τα καλά της λόγια. Σημεριζόμεθα κάποια σχόλια που έγιναν εις ό,τι αφορά την ενδυνάμωση της ε, ψηφιακής ε, διάστασης μείωσης της ψηφιακής διαίρεσης, η ενδυνάμωση των κέντρων είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης για τον εθισμό, τον ψηφιακό εθισμό. Ε, δεν είναι αυτό το πρόγραμμα που θα το καλύψει αυτό, αλλά έχουμε άλλα προγράμματα που καλύπτουν αυτό το θέμα. Συνολικά σας πρέπει να πω ότι ήταν ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας και σας ευχαριστώ. Τώρα, η εισηγήτρια για ένα τελευταίο σχόλιο. Η κυρία Μίλναρ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Λίγος πολύ ευθυγραμμίζονται με τη συζήτηση που είχαμε κάνει ως κοιόδης. Σας ενημερώνω ότι Εξετάζομαι λύσεις που θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ε, όπως γίνεται στην κοινή επιχείρηση και σε άλλα προγράμματα ε, όπως στο Συνδέοντα στην Ευρώπη. Επίσης θέλουμε μια συμβιβαστική λύση για να ανοίξει το πρόγραμμα σε τρίτες χώρες για την τεχνητή νοημοσύνη. Εξετάσαμε την πρόταση της Κομισιόν για, και περιμένουμε το πλαίσιο που θα δώσει δεοντολογική καθοδήγηση χωρίς να υπονομεύεται η καινοτομία. Για την ψηφιακή διαίρεση πιστεύουμε στην προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου προγράμματος και πρέπει να οικοδομήσουμε ικανότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όχι να ωφεληθούν μόνο οι πιο προηγμένες χώρες και τα ψηφιακά κέντρα όπως ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Ε, θα πρέπει να είναι ένα δίκτυο που μπορεί να διανύμει και να ενδυναμώνει σε περιφερειακό επίπεδο ε, τους στόχους μας και να τους επιδιώκει όπως είπε και η συνάδελφος Γκρίφιν. Για τον ψηφιακό γραμματισμό πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι κομμάτι αυτού του προγράμματος, δεν νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί γιατί απλώς δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια. Μιλάμε για 9,2 δις ευρώ, αυτός είναι ο προϋπολογισμός και δεν πρέπει να τον παραφορτώνουμε γιατί αλλιώς θα είναι υπερβολικά πολλοί οι στόχοι και στο τέλος δεν θα επιτευχθούν. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Αμλίναρ και ένα προσωπικό σχόλιο. Όλη μου τη ζωή ασχολήθηκα με τον κλάδο τεχνολογίας πληροφοριών και ευχαριστώ ε, την ε, για την συνεισφορά σας. Έχω εμπειρία από μεγάλους υπολογιστές, PC, το διαδίκτυο και ελπίζω ότι από αυτή την πρωτοβουλία θα βγει κάτι πολύ χρήσιμο. Να σας πω ότι η ψηφορία στην Ήτρα θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου. Και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η νέα χρήση πληροφοριών στον δημόσιο τομέα. Αναδιατύπωση. Σας υπενθυμίζω ότι η παρούσα πρόταση είναι αναδιατύπωση και ότι ε, ισχύουν ειδικοί κανόνες όταν κατατίθενται τροπολογίες. Είναι το άρθρο 104. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι τροπολογίες γίνονται δεκτές μόνο αν αφορούν εκείνα τα μέρη της πρότασης που, αφορά, που περιέχει συγγνώμη, αλλαγές τροπολογίες σε μέρη τη πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα μπορεί να γίνουν μόνο κατά εξαίρεση και κατά περίπτωση. Μόνο έτσι μπορεί να γίνουν δεκτές από τον ή την πρόεδρο εάν θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο για ε, ε, επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες προς άλλες τροπολογίες που είναι παραδεκτές. Τέτοια οι λόγοι θα πρέπει να αναφέρονται σε γραπτή αιτιολόγηση προς τις τροπολογίες. Κατόπιν τούτου θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σίλη Κιώτη, για την παρέμβασή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές της εκθεσής, καθώς και τους συνεργάτες τους, για τις επικοδομητικές συναντήσεις που είχαμε μέχρι σήμερα, Είμαι σίγουρος πως παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν σε επιμέρους θέματα, ο στόχος είναι κοινό και με συλλογική δουλειά θα επιτύχουμε τη βελτίωση του κειμένου στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ε, η πρόταση της Κομισιόν είναι μια πολύ καλή βάση για συζήτηση της αναθεώρησης, αναδιατύπωσης οδηγίας και όπως πολύ ορθά ε, αναφέρατε Πρόεδρε, αυτό αφορά εκείνα τα, ε, εκείνες τις πρόνοιες ακριβώς που αναδιατυπώνονται και ε, εκεί πρέπει να εστιαστούν και οι όποιες τροπολογίες. Ε, ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι το Ευρωκοινοβούλιο στο μόνο εκλεγμένο σώμα οφείλει να προωθήσει και νέες προτάσεις, εστιάζοντας περισσότερο στις ανάγκες της κοινωνίας. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ένα θεμελιώδης ανθρώπινο δικαίωμα. Θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε πως τα ανοιχτά δεδομένα θα αποφέρουν πραγματικό όφελο στην κοινωνία και των ανθρώπων και θα αξιοποιούνται όχι μόνο από τις μεγάλες εταιρείε που έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά κυρίως και για την ενδυνάμεση των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει, κατά την άποψή μου, τα δεδομένα να δίνονται δωρεάν, όπου είναι δυνατόν, και όταν απαιτείται επιβολή τελών να περιορίζεται στο οριακό κόστος. Σε όλε ανεξέλεκτε όμω τι περιπτώσει και για όλα τα δεδομένα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμό τη Ένωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπω εγκρίθηκε πριν από λίγου μήνε. Εξίσου σημαντικό είναι να συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση τη Κομισιό ε, και ο αντίκτυπο που θα έχει η εν λόγω οδηγία στην αγορά εργασία. Ε, δηλαδή στι υφιστάμενε θέσει εργασία αλλά και σε ώστε να διασφαλίσουμε τη δημιουργία νέων ποιοτικών και αξιοπρεπών εργασία. Για να επιτύχουμε την υλοποίηση τη αναθεωρημένη οδηγία, είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη και οι φορεί του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα οι μικρέ τοπικέ κοινότητε και τα κράτη που πλήττονται από την οικονομική κρίση, να στηριχτούν οικονομικά από την Ένωση, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια στι απαιτήσει τη οδηγία και να διαθέτουν με αποτελεσματικό, γρήγορο και εύκολο τρόπο όλε τι πληροφορίε. Όσον αφορά τα δεδομένα υψηλή αξία, θεωρούμε πω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ενισχυμένο ρόλο στη διαμόρφωση του καταλόγου των ε, συνόλων δεδομένων υψηλή αξία. Γι' αυτό και προτείνουμε να διατηρηθεί το Delegate Act, η πράξη κατεξιοδότηση, αντί να πάμε σε Implementing Act, εκτελεστική πράξη. Ε, και εδώ θεωρώ ότι το σύνολο των ε, σκιώδων συμφωνεί με αυτή τη θέση αλλά και να προταθεί εξ αρχή ένα κατάλογο, ο οποίο να αξιοποιηθεί ω βάση και να οκληρωθεί από την Κομισιόν, αφού βέβαια προηγηθεί διαβούλευση, ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψει όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Κλείνοντα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημαντικό θέμα, για το οποίο υπάρχει διάσταση απόψεων. Τι δημόσιε επιχειρήσει και τη συμπερίληψή του ή όχι στο πεδίο εφαρμογή τη εν λόγω οδηγία. Κατά την άποψή μα, η προτινόμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογή στι δημόσιε επιχειρήσει, ώστε και σε εθελοντική βάση, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρέ στρεβλώσει με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να ενταθούν ακόμα περισσότερο οι άνισοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων επιχειρήσεων στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν και ανταγωνίζονται στο ίδιο πεδίο, στην ίδια αναγορά. Οι ιδιωτικέ επιχειρήσει θα υποφελούνται από τι πληροφορίε που θα του δίνονται από τι δημόσιε επιχειρήσει, καθώ θα αξιοποιούν τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν με δημόσιο χρήμα για να βελτιώνουν τι υπηρεσίε του και να υπερισχύουν στην αγορά, αυξάνοντα τα κέρδη του. Δηλαδή, παρόλο που οι ιδιωτικέ επιχειρήσει δεν θα είναι υποχρεωμένε να παρέχουν καμιά πληροφορία, θα παίρνουν τα δεδομένα που θα δίνουν οι δημόσιε επιχειρήσει και θα τι ανταγωνίζονται από θέση ενισχύω. Έτσι, οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν ελάχιστες πιθανότητες να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό, ενώ δεν αποκλείεται να υποχρεωθούν να προχωρήσουν και σε αύξηση της τιμής του κόστου για την προσφερόμενη υπηρεσία τους προκειμένου να επιβιώσουν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να διατηρήσουμε τις δημόσιες επιχειρήσεις εκτός του πεδίου εφαρμογή αυτής της οδηγίας, όπως ήταν μέχρι σήμερα. Ζητάμε δηλαδή η απόφαση σχετικά με το αν επιτρέπεται ή όχι περαιτέρω χρήση των πληροφοριών και υπό ποιε συνθήκε να αποφασίζεται αποκλειστικά από τι ίδιε τι δημόσιε επιχειρήσει. Ωστόσο, εάν η πλειοψηφία επιθυμεί να διατηρηθούν οι αναφορέ στι δημόσιε επιχειρήσει, τότε θεωρώ πω πρέπει να συμπεριλάβουμε οπωσδήποτε σχετική αναφορά και στι ιδιωτικέ επιχειρήσει, οι οποίε θα παρέχουν τι ίδιε υπηρεσίε γενικού συμφέροντο μέσω σύμβαση, μέσω ενό συμβολίου που θα υπογράφουν με οργανισμό του δημόσιου τομέα. Δηλαδή εκεί που δραστηριοποιούνται στον ίδιο ε, τομέα θα πρέπει και οι ιδιωτικέ επιχειρήσει να αποχρώνονται να δίνουν τις πληροφορίε αυτές για να μην δημιουργείται ε, μια αδικία, μια ανισότητα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. And now... Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για το ΕΛΚ. Ο κύριος Μπόνι. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω τον εισηγητή πρώτα απ' όλα για την ε, συνεκτική ε, έκθεση. Η οδηγία αυτή είναι βήμα μπροστά στη διεύρυνση της χρήσης των πληροφοριών του δημοσίου τομέα ε, στα πλαίσια της οικονομίας των δεδομένων. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους φορείς του δημοσίου τομέα να διαθέτουν δημόσια δεδομένα το ταχύτερο δυνατόν, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή. Αυτό θα ήταν χρησιμότατο μέσα από διεπαφές εφαρμογών και προγραμμάτων και να διευκρινίσουν την ανάκτηση του κόστους ε, ανωνυμοποιημένων δεδομένων ως προϋπόθεση για τη νέα ε, ε, χρήση με πλήρη σεβασμό, του σεβασμού στα δεδομένα. Η αναδιατύπωση λαμβάνει υπόψη δεδομένα από δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις γενικού ε, ενδιαφέροντος ε, και άλλων που βρίσκονται εκτός του ε, δημοσίου τομέα, όμως εκεί όπου υπάρχει μεγάλος έλεγχος κρατικός. Πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις δημόσιες αυτές επιχειρήσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια, βασική, μια βάση για καλές πολιτικές δεδομένων στο μέλλον. Η διαδικασία όμως θα πρέπει να σέβεται τις αρχές του θεμητού ανταγωνισμού. Το είπε και ο εισηγητής. Θα πρέπει όλοι να υπόκεινται στις ίδιες διαδικαστικές προϋποθέσεις χωρίς διάκριση μεταξύ δημοσίου ιδιωτικού. Ε, δεν υπάρχει ε, λόγος για διακριτική μεταχείριση. Ναι, λοιπόν, ε, να είναι ε, βασικός εταίρος οι δημόσιες επιχειρήσεις, αλλά να σέβονται ε, συγκεκριμένες αξίες. αξία αξίας ε, σειρέ δεδομένων, αυτό είναι σημαντικό, ε, σημαντικός στόχος. Θα πρέπει να έχουμε κατάλογο και κατηγορίες σειρών δεδομένων για να έχουμε εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε εδώ κινητικότητα, μεταφορά δεδομένων, στατιστικές, ειδικά δεδομένα, ε, παρατήρηση, ε, ε, παρατηρήσεις GPS, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια δεδομένα θα είναι δωρεάν, αναγνώσιμα, προσπελάσιμα για να μπορούν να κατεβαίνουν. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποιο μοντέλο είναι καλύτερο, ε, ποιο μοντέλο είναι καλύτερο ε, να δούμε τις κατεξουσιοδότηση έναντι των ε, εκτελεστικών πράξεων. Οι νέε προϋποθέσεις και διατάξεις για την προσπελασιμότητα θα πρέπει να εγγυώνται την νέα χρήση και να είναι και διαλειτουργικά, διότι θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να διαδώσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Και τέλος το πεδίο εφαρμογής, το εύρος της οδηγίας ε, για τις ε, δημόσιες ε, υπηρεσίες δεν πρέπει να καλύπτει εκείνες τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό των ειδικών υπηρεσιών με βάση την οδηγία για την προστασία δεδομένων. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες και ειδικές προϋποθέσεις ασφαλείας θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι είναι δυνατόν και πότε χρειάζονται πρόσθετες ε, προϋποθέσεις ε, για να, για να κάνουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ των ε, επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπόνη. Και τώρα για, σοσιαλ, για τους σοσιαλιστές... Α, ο κύριος Σορίνιο πάλι για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας πω ότι εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό κείμενο και το έχουμε ξανασυζητήσει. Τα δεδομένα είναι θεμελιώδους σημασίας εδώ και θα πρέπει να είναι συμβατά με τις ανάγκες ασφαλείας και προστασίας των πολιτών. Ε, θα πρέπει να δούμε τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και τι πρόσβαση θα έχουν ε, και οι δύο έχουν, είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των δεδομένων αλλά και θα πρέπει να δούμε την πρόσβαση στους παρόχους και πώς γίνεται η διαχείριση. Η τάση είναι να έχουμε ε, δημόσια πρόσβαση στα δεδομένα με βάση ε, ελεύθερη και ουδέτερη σε ό,τι αφορά ε, τα γεωγραφικά δεδομένα. Αυτά θα πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ. Και τώρα έχουμε επιπλέον μια ευκαιρία να ξαναδούμε και να μοιραστούμε την έννοια την ενός ευρωπαϊκού δικτύου δημοσίων ε, υπηρεσιών. Ε, με το 5G και τα άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. E um, από, από την ομάδα ECR, ντρέπομαι να πω ότι δεν υπάρχει συμμετοχή για να μιλήσει κανείς, άρα θα μιλήσει για τους φιλελευθέρους ο κύριος Πέτερσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι σύντομος γιατί συμφωνώ με τους προλαλήσαντες σε γενικές γραμμές με όλα όσα είπαν. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Σιλικιώτη για την πολύ καλή συνεργασία και για την καλή του δουλειά ε, στο ε, σχέδιο έκθεσης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ σημαντική για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας των δεδομένων στην Ευρώπη και πιστεύουμε ότι υπάρχει πολύ καλή, πολύ ε, καλή συλλογιστική πίσω από την εναρμόνιση Και βεβαίως ε, η πρόσβαση σε δυναμικά δεδομένα και σε υψηλής, ε, σε μεγάλης αξίας ε, δημόσια δεδομένα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό στην προσπάθειά μας αυτή. Μπορεί να υπάρχουν συμφωνίες αποκλειστικότητας μεταξύ δημοσίων φορέων και ιδιωτικών φορέων και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Όλα αυτά νομίζω καθιστούν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το νομοθέτημα. Ο εισηγητής εισάγει νέα στοιχεία στο σχέδιο έκθεσης για μας στην ομάδα ε, των φιλελευθέρων θα προτιμούσαμε οι δημόσιες επιχειρήσεις να είναι στο πλαίσιο της οδηγίας όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ε, έχουμε την πρόθεση να συζητήσουμε περισσότερο όσον αφορά τη συμπερίληψη των συνόλων δεδομένων ε, μεγάλης αξίας με αυτέ τι παρατηρήσεις κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι εναγωνίω αναμένουμε περαιτέρω συνεργασία για την ολοκλήρωση αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πίτερσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης σε ένα πολύ σημαντικό φάκελο για μας Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά έκανε σημαντικό βήμα μπροστά, εισάγοντας αυτήν την έννοια των σειρών των δεδομένων ε, υψηλής αξίας. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον και είναι τόσο σημαντικό. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε μια κατάσταση όπου έχουμε χαρτογραφικά δεδομένα, τα οποία παρέχονται με αμοιβή στην Google, ας πούμε, που μπορεί να πληρώσει. Ε, ενώ και αυτό χρησιμοποιείται για να βελτιωθούν τα δεδομένα. Αλλά προγράμματα όπως Open Street Maps, οι μικροί ανταγωνιστέ, προγράμματα των πολιτών δεν έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Και η Κομισιόν είδε στην ε, ανάλυση αντικτύπου ότι το κόστος χρέωσης για, αυτά, για αυτές τις σειρές ε, υψηλής αξίας δεδομένων ξεπερνούν τα ε, Είναι σημαντικό να είμαστε πολύ φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά αυτές τις σειρές δεδομένων υψηλής αξίας και θέλω με την προσέγγιση να έχουμε ένα παράρτημα που καταγράφει κατηγορίες ε, σειρών δεδομένων υψηλής αξίας που, πρέπει, που θα είναι προσπελάσιμα σε όλους. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πραγματικό βήμα μπροστά έναντι της πρότασης της Κομισιόν που προτείνει να ορίζει μόνο η Κομισιόν μέσα από κατεξουσιοδότηση πράξη τα δεδομένα αυτά, αυτό πάει πάρα πολύ. Και δίνει μεγάλη διακριτική ευχέρεια στην Κομισιόν. Εμείς πρέπει ως νομοθέτης να αναλάβουμε σοβαρά το ρόλο μας, να ορίσουμε αυτές τις σειρές δεδομένων υψηλής αξίας. Όμως πρέπει να υπάρχει κατεξουσιοδότηση πράξη για να τροποποιείται αυτός ο κατάλογος στο μέλλον, γιατί μπορεί να υπάρξουν και εξελίξεις στο μέλλον. Και μια κατεξουσιοδότηση πράξη θα δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να ελέγχει αυτή τη διαδικασία από ότι η εκτελεστική πράξη. Γι' αυτό προτιμούμε την πρώτη προσέγγιση. Γενικά είμαστε πολύ ευτυχείς από την προσέγγιση που ακολουθεί ο εισηγητής. Θέλουμε όμως να επισημάνουμε και δύο προβλήματα. Το ένα αναφέρθηκε ήδη από συναδέλφους. Πιστεύουμε ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής. Πρώτον, για το λόγο ότι έχουν τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα δεδομένα. Αν δούμε τις δημόσιες επιχειρήσεις, τον κοινή ωφέλεια, τις μεταφορές, αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία τεράστια για την κοινωνία ευρύτερα και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Επίσης θέλουμε να φροντίσουμε παράλληλα ότι αυτό δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτό ε, γίνεται, ε, υπάρχει στην πρόταση της Κομισιόν. Να το ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο. Να συμπεριλάβουμε και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ε, κάνουν, προσφέρουν υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος που μοιάζουν με τις δημόσιες επιχειρήσεις για να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουν την ίδια μεταχείριση αλλά η συμπερίληψη δημοσίων επιχειρήσεων για μας είναι πολύ σημαντική. Δεύτερο σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ προσεκτικά αξιολόγησε τα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν στο δημόσιο τομέα από, ε, με βάση την οδηγία ε, για τη βάση δεδομένων. Δηλαδή κάποιο που θέλει να ξαναχρησιμοποιήσει ανοιχτά δεδομένα να μην μπορεί να συνδυάζει δεδομένα ε, από διάφορες πηγές γιατί οι προϋποθέσεις είναι διαφορετικές. Εκεί καλό είναι να κρατήσουμε την πρόταση της Κομισιόν ότι δεν πρέπει να ασκούν οι δημόσιες επιχειρήσεις το δικαίωμα της βάσης δεδομένων. Κατά τα άλλα είμαστε ευτυχείς με την έκθεση και προσβλέπουμε και σε συνεργασία από εδώ και πέρα. Ε, Ευχαριστώ κυρία Ρέντερ. Ευχαριστώ κυρία Ρέντα. Σκιώδης άλλος δεν υπάρχει. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Ε, πολύ. Προφανώ ο δημόσιο τομέα έχει πάρα πολλά δεδομένα στη διάθεσή του γεωγραφική, μετεωρολογική, εκπαιδευτική φύσεω, οικονομική, κοινωνική. Συνεπώ, είναι μία ε, πηγή ανάπτυξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον τομέα ε, Τη τεχνική νομοαιμοσύνης ή βελτίωση της αποτελεσματικότητας ε, της ε, δημόσιας πολιτικής. Υπάρχουν στοιχεία για την ασφάλεια, για τις μεταφορές. Είναι σημαντικό λοιπόν να συμπεριληφθούν οι δημόσιες υπηρεσίες στο πεδίο εφαρμογή. Όμως ε, υπάρχει μια μικρή αντίρρηση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην, για την κατάσταση των δημοσίων υπηρεσιών ε, που πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες ε, γενικής ε, οικονομικής ωφέλειας γιατί είναι σε ένα επίπεδο, σε ένα πλαίσιο ανταγωνιστικό και δεν πρέπει να βρίσκονται σε μια μειονεκτική θέση. Υπάρχουν όμως πληροφορίες οι οποίες είναι, υπάρχουν πληροφορίες που είναι ε, πολύ σημαντικές, ανταγωνιστικές και δεν πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ε, αντιπάλων. Γι' αυτό ακριβώς ε, δεν πρέπει να υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού με, με, υπηρεσίες οι οποίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής. Πρέπει αυτές οι υπηρεσίες να μπορούν να καθορίσουν τις, τους όρους χρήσης των ίδιων των δεδομένων τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση, τις παρατηρήσεις του και θέλω να πω ότι είναι καταπληκτικό τι θησαυρό δεδομένων έχουμε στις δημόσιες διοικήσεις που μπορούμε να διαθέσουμε στους πολίτες μας. Υπάρχει μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό, κυρίως για τις ΜΜΕ εδώ. Όμως και μια κριτική παρατήρηση. Και συμφωνώ με την συνάδελφο Γκροστέτ εδώ. Δεν πρέπει να ε, το παρακάνουμε και να χάσουμε τα ωφέλη που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση από, αυτή, αυτό και να επιβάλλουμε σε όλες τις διοικήσεις τι δεδομένα από ποια ημερομηνία και μετά πρέπει να διαθέτουν. Αυτό θα είναι μεγάλο, μεγάλος φόρτος για τις δημόσιες διοικήσεις. Υπάρχουν δε και ευαίσθητα δεδομένα ε, για τις συγκοινωνίες σε μια πόλη, τις μεταφορές, ε, οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για να αποφεύγουμε μποτιλιαρίσματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς που άπτονται της ασφάλεια. Γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτική σε σχέση με την υποχρεωτική διάθεση δεδομένων ε, από την χ ημερομηνία από τις δημόσιες ε, διοικήσεις. Παρακαλώ να το ξαναδούμε αυτό Μήπως μπορούμε να το περιορίσουμε λιγάκι. Όπως και η κυρία Γκροστέτ, ε, νομίζω ότι οι δημόσιες ε, επιχειρήσεις που είναι ανταγωνιστικές ε, τρίτες, εκεί θα πρέπει να ισχύσουν άλλα κριτήρια αξιολόγησης, άλλα μέτρα και σταθμά και τέλος ε, εδώ θα καταθέσουμε τροπολογία ε, για το θέμα της ευθύνης και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ε, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε το δημόσιο να διαθέτει δεδομένα και αν υπάρξει πρόβλημα με τα δεδομένα αυτά και δημιουργηθούν από τις εφαρμογές ζημίες δεν μπορούμε να ε, θεωρήσουμε ότι υπεύθυνε είναι οι δημόσιες υπηρεσίες που τα διέθεσαν. Το θέμα δηλαδή της ε, ευθύνη θα πρέπει να το δούμε. Χαίρομαι για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα και ας δούμε λίγο σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής αν αυτό το ευρύ πεδίο όπως προβλέπετε και όπως ε, παρουσιάστηκε ε, και από τον εισηγητή και από συναδέλφους μήπως μπορεί αυτός ο το, ευρύ, το ευρύ πεδίο εφαρμογής μπορεί να περιοριστεί λιγάκι. Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ, κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον 21ο αιώνα τα δεδομένα έχουν οικονομική αξία, σαφές. Άρα καλωσορίζουμε την οδηγία η οποία δημιουργεί δυνατότητα περαιτέρω χρήσης. Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ε, όμως και ένα νομοθετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των δεδομένων, για την οικονομία, για την εργασία. Θα πρέπει να δούμε όμως ε, αυτά τα ε, δεδομένα είναι ένα παραπροϊόν που μπορεί να αξιοποιηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί ή είναι βασική πρώτη ύλη που θα πρέπει να ειδωθεί και να ε, αξιολογηθεί διαφορετικά. Είναι οικονομικό αγαθό τα δεδομένα ε, των 21ο αιώνα που βρίσκονται και στα χέρια δημοσίων επιχειρήσεων. Ε, υπάρχουν υπηρεσίες που είναι δημόσιες αλλά ανταγωνίζονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και η περαιτέρω ε, χρησιμοποίηση από αυτές θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά εις ό,τι αφορά την λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται. Πολλές φορές ε, τα δεδομένα συνδέονται με κόστος και ε, αν η ε, οι επικερδείς ε, διοχετευτούν στις ιδιωτικές υπηρεσίες ενώ οι λιγότερο επικερδείς μείνουν στο δημόσιο, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Και επίσης πρέπει να δούμε και τους φορολογούμενους, γιατί πολλές φορές οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν μεγάλες δαπάνες, αλλά δεν έχουν ε, κέρδη υψηλά. Και σε κάποιες περιπτώσεις και μέσα από αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για στρέβλωση του ανταγωνισμού. Επίσης, αν η πρόθεσή μα είναι να υπάρχει ασφάλεια δικαίου με την οδηγία, τότε ο οδηγό. Ε, ο ορισμός συγγνώμη, των ε, σειρών δεδομένων υψηλής ε, αξίας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που προτείνεται από την Κομισιόν και τη σχετική πράξη. Χρειάζεται δημοκρατικός έλεγχος, ούτως ώστε να μην βρεθούμε προ δυσαρέστων εκπλήσεων, εκπλήξεων όταν μπορεί να ορίζει κατά το δοκούν η Κομισιόν τις σειρές δεδομένων υψηλής αξίας. Ευχαριστώ. Και τώρα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης, όπως επίσης και τους ευρωβουλευτές για τα σχόλια τους. Η έκθεση αναγνωρίζει με πολύ ωραίο τρόπο την αξία των δεδομένων αυτών ε, και για τους πολίτες ε, και για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Η υποστηρίζει τη χρήση των ε, υψηλής αξίας ε, συνόλων δεδομένων που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά καταλαβαίνουμε και την ανάγκη πλαισίωση σε αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα κάνει σε μια πρώτη φάση. Προστασία δεδομένων αναφέρθηκε. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η οδηγία θα ισχύσει με πλήρη σεβασμό των κανόνων προστασίας δεδομένων. Όσον αφορά τη χρέωση, τα τέλη για την ε, εκ νέου χρήση των δεδομένων είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια της αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ε, αναδιόμενες επιχειρήσεις. Ε, οι τεχνολογικοί γίγαντες μπορούν να πληρώσουν τα τέλη αυτά σε κάποιες δημόσιες επιχειρήσεις. Όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνει ότι το τέλος είναι ένα κλάσμα μόνο ε, του ωφέλους που μπορεί να υπάρχει το άνοιγμα αυτό των δεδομένων. Μιλάμε για τομείς, για ενέργεια, νερό, ε, μεταφορές, όπου υπάρχουν πολλά δεδομένα και υπάρχουν και προβλήματα που έχουν επισημανθεί. Έχουμε πάρα πολύ προσεκτικά δει την ανταγωνιστική θέση των δημοσίων επιχειρήσεων υπό το φως οποιονδήποτε ενδεχομένων μέτρων και πιστεύουμε ότι οι περιορισμένες υποχρεώσεις που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια εξισορροπημένη λύση. Δεν μιλάμε για ανοιχτά δεδομένα για τις δημόσιες επιχειρήσεις, σε καμία περίπτωση. Μια τελευταία ε, παρατήρηση, να το συνδέσω με αυτό που συζητήθηκε προηγουμένως, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Υπάρχουν δυνατότητες στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη, χρηματοδότησης κάποιων ε, δραστηριοτήτων από πλευράς κρατών μελών. Όσα κράτη-μέλη έχουν ε, ζητήσει να συμμετέχουν. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος λέει, ο κύριος Σίλικιώτης για τα τελικά του σχόλια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδελφούς ε, για τις παρεμβάσεις τους και για τις παρατηρήσεις τους. Ε, ε, δεν θα επαναλάβω ζητήματα που τέθηκαν εδώ. τα μόνα σημεία που θέλω να θίξω ξανά είναι το θέμα της ότι πρέπει να είναι πράξη κατεξιοδότηση, όχι εκτελεστική πράξη, για να μπορεί να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία και ε, να είναι σωστό να κατευθεί ένα κατάλογος ε, για του τομεί ιδιαίτερα για τα δεδομένα υψηλή αξία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι δημόσιες επιχειρήσει, ε, καταλαβαίνω τη σημασία και που το έθεσαν πολλοί συναδέλφοι, όμω. συμφωνώ με του συναδέλφου που έθεσαν και το θέμα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε συνθήκε αθέμητη ανταγωνισμού. υπάρχουν πάρα πολλοί δημόσιες επιχειρήσεις, ειδικότερα που είναι σε ε, ε, ε, δήμους, σε κοινότητες, σε τομείς που υπάρχει έντονος ανταγωνισμός ιδιωτικές επιχειρήσεις και γι' αυτό δεν πρέπει να οδηγήσουμε τα πράγματα σε ένα θέμα των ανταγωνισμών. Είναι γι' αυτό που στην αρχική εισήγηση έθεσα και τη θέση ότι θα μπορούσε να βρούμε τρόπον εκεί που υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν συμβόλαια με το κράτος, που κάνουν ε, δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα, ε, να υποχρώνουν και εκείνοι να παρέχουν κάποια δεδομένα. Άρα αυτό το θέμα των δημόσιων επιχειρήσεων, επειδή κυρίω είναι επιχειρήσει σε οργανισμού κοινή ωφελία, είναι οργανισμοί κοινή ωφελία, ε, χρειάζεται ε, ακριβώ πολύ προσοχή και θεωρώ και πιστεύω ότι μαζί με τους κοινού εισηγητές και μετά με ολόκληρη την Επιτροπή θα βρούμε ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να με θέσουμε τις δημόσιες επιχειρήσεις ε, σε μειονεκτική θέση. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ε, ε, αναμένω ότι αυτή η συζήτηση και η συνεργασία μας θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες ώστε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για την επαναδιατύπωση της οδηγίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι η προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών για το σχέδιο έκθεσης έχει οριστεί για τις 11 Οκτωβρίου 2018. 11 Οκτωβρίου 2018 ε, είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, το Ταμείο Άμυνα, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θέσπιση του, θα, τη σύστασή του μάλλον, θα ήθελα να σα πω ότι είναι ένα νέο πρόγραμμα που, που συνδυάζει την έρευνα και την βιομηχανική καινοτομία για αμυντικούς σκοπούς είναι ένα ε, ταμείο υπό ε, το ορίζον ε, Ευρώπη 13, 13 δις προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4,1 εξ αυτών θα δοθούν στην, σε προγράμματα ανταγωνιστικά έρευνας και καινοτομίας είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πρόγραμμα και από απόψεως χρηματοδοτικής και από απόψε Εμβέλεια. Έχουμε λάβει για την ώρα 457 τροπολογίες ε, επί της πρότασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 98 από τον εισηγητή ε, στο σχέδιο έκθεσής του. Έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας για την εξέταση του θέματος αυτού και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μας, τον εισηγητή, τον καθηγητή Κρασνοντέμσκι, ο οποίος θα παρουσιάσει τις τροπολογίες εντός 5 λεπτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, πολλές οι τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που κατέθεσαν 357 τροπολογίες ε, βάσει των οποίων μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι δεν συμφωνούμε όλοι ως προς το ταμείο αυτό. Ένας από τους στόχους είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του μυντικού τομέα στην Ευρώπη, αλλά Στη μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τις γεωπολιτικές αλλαγές που συμβαίνουν ε, στον περιβάλλοντα χώρο της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες, αλλά υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες εκφράζουν κάποια δυσαρέσκεια, κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα κινείται προς την στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και υπάρχουν ανησυχίες ε, ότι μπορεί να περιοριστούν τα προνόμια των κρατών μελών ε, στον αμυντικό τομέα. Όμως, Κάποιε άλλε χώρε, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες από το Ταμείο αυτό. Θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία από πλευρά ευρωπαϊκή Ένωσης να επιτύχει μια στρατηγική αυτονομία στόχοι όπως η μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής άμυνας, το να καταστεί η Ευρώπη ανεξάρτητη από προϊόντα τρίτων χωρών. Ένας ακόμη στόχος είναι η προώθηση της καινοτομίας. Συνεπώς υπάρχουν τροπολογίες που σκοπό έχουν την αύξηση των κονδυλίων για επαναστατικές τεχνολογίες. Όλες αυτές οι τροπολογίες είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτες. Υπάρχουν κάποια ζητήματα με το άρθρο 7 και το άρθρο 8. Συμφωνούμε ότι πρέπει να τελειοποιηθεί, πρέπει να τελειοποιηθούν τα άρθρα αυτά, αλλά είναι διαφορετικές ιδέες σε σχέση με το πώς πρέπει να γίνει αυτό. Θα δουλέψουμε με σκοπό το συμβιβασμό για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια δικαίου για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις αλλά και για, το, για, την, για, την προάσπιση των συμφερόντων στα οποία αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα ακόμη ζήτημα. Σύμφωνα με το άρθρο 10, οι φορείς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τους φορείς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που λένε ευρωπαϊκό χρήμα για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε σε αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια πιο... ένας πιο περιεκτικός ορισμός του τι θα πει η ευρωπαϊκή ε, επιχείρηση. Νομίζω ότι γίνεται μια αρκετά ρεαλιστική αξιολόγηση του τι εννοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, την, με το πρόγραμμα αυτό που σκοπό έχει να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Άμυνα και ελπίζω τη συμμετοχή των, ε, των φορέων που πληρούν τα κριτήρια θα είναι η κατάλληλη. Τώρα για χώρες ε, εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τρίτε χώρες, θα ισχύσουν διαφορετικά κριτήρια. Το κοινό έδαφος είναι αρκετά εκτεταμένο, νομίζω ότι φάνηκε αυτό και στι συναντήσει των ε, σκιωδών έχουμε πιθανότητες να καταλήξουμε σε έναν καλό συμβιβασμό Να ευχαριστήσω την κυρία Γκροστέτ για την ε, συνεργασία της. Ελπίζω να τα καταφέρουμε γιατί δεν, έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκροστέτ για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, που ήταν άλλωστε απαραίτητη, μια και πρόκειται ε, για ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Ωστόσο, τον ευχαριστώ τον συνάδελφο για την στάση του και τη συνεργασία που είχαμε. Το Ταμείο αυτό 2021-2027 είναι σημαντικό ε, όσον αφορά τα στοιχεία που αφορούν την οικοδόμηση ικανότητας ε, και την ε, έρευνα. Ο προϋπολογισμός είναι 13 δις και είναι πολύ σημαντικό αυτό και άλλωστε υπόθηκε οπωσδήποτε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τρόπο αποτελεσματικό και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμιστεί η αριστεία και η ανταγωνιστικότητα στη διάρκεια της και στη φάση της επιλογής των ε, προγραμμάτων. Άλλωστε αυτό υπογραμμίζεται και στις τροπολογίες. Οπωσδήποτε πρέπει να, ε, να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε ε, χωρίς λόγο καινούργιες διαδικασίες Ε, και ε, έχουμε δυστυχώς πλήστα όσα παραδείγματα. Χρειαζόμαστε ευελιξία στην υλοποίηση εάν θέλουμε να ε, συλλέξουμε όσο γίνεται περισσότερα προγράμματα. Αυτό το ταμείο παρά το πρώτο πρόγραμμα 19-20 είναι καινοτομία, είναι νεοτερισμός μάλλον για την Ευρώπη. Πρέπει να δούμε τις υπάρχουσες ε, καταστάσεις, να δούμε εάν ε, καλύπτονται οι απαιτήσει του Ταμείου και θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε νέες συνεργασίες. Ε, σε αυτό το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Αριστείας θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τα καλύτερα project σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα στο πρόγραμμα 19-20 και το Ταμείο μέχρι το 27 θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ειδικέ δράσεις της πτυχής έρευνας που θα ακολουθήσει την πτυχή ανάπτυξη. Μαζί με άλλους συναδέλφους του ΕΡΛΚ προτείνουμε εναρμόνιση των διαδικασιών ε, σε σχέση με την ε, ε, διανοητική ιδιοκτησία των δύο πτυχών γιατί θεωρώ ότι είναι πιο λογικό. Τέλος, και αυτός άλλωστε είναι και ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτού του Ταμείου, θα πρέπει να επαγρυπνήσουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εξαρτάται πλέον και σε βάθος χρόνου από εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα. Έχουμε υποβάλει λοιπόν ε, πολλές τροπολογίες σχετικά με τα κριτήρια ε, ε, διανομής και με τις επιλέξιμες οντότητες και τον τρόπο επιλογής. Πρέπει να επαγρυπνήσουμε για τα χρήματα και να προστατεύουμε τα χρήματα των ε, ε, φορολογουμένων πολιτών αλλά και να υπαγρυπνούμε γενικά γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αποθαλμιούν την ε, Ευρώπη. Αυτά και ευχαριστώ τον εισηγητή και είμαι βεβαία ότι θα συνεργαστούμε θετικά έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα, μια έκθεση πολύ φιλόδοξη. Ευχαριστώ πολύ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες η κυρία Γκρίφιν, η οποία αντικαθιστά τον κύριο Μαρτάν, νομίζω, ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Εντουάρ λυπάται, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει ο ίδιος. Ε, ανέλαβε μετά από την τιμωρία του. Ε, έχω τη δυνατότητα να Είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε προηγουμένως τη θέση του. Τώρα όμως άρχισαν οι συναντήσεις των σκιωδών και πρέπει να μιλήσουμε για κάποια επιχειρήματα. Για την επιλεξιμότητα η συμβαστική λύση θεωρείται ε, ε, το, κατόφλι. Ε, όμως ε, τώρα θα πρέπει να δούμε και τις βιομηχανικές δυνατότητες στα κράτη-μέλη που κάνουν ε, έχουν εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες. Ε, ε, θα πρέπει να καλυφθούν εξαρτήσεις και βιομηχανικά κενά. Αν δεν το κάνουμε αυτό και αν σε 7 χρόνια βρεθούμε ακριβώς στην ίδια είχε και χειρότερη θέση, με την εξάρτηση που έχουμε στην... Ε, θα έχουμε εξάρτηση, αυξήσει την εξάρτηση από την Αμερική και την Κίνα. Πού είναι η στρατηγική μας αυτονομία. Για τη δεοντολογία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνονται δεοντολογικοί ε, εκ των προτέρων έλεγχοι και θα πρέπει να γίνονται και μετά από κοινοβουλευτικό αίτημα το περιεχόμενο είναι πολλές φορές ε, ε, διαβαθμισμένο, αλλά δεν μπορούμε παρόλα αυτά να μην το λάβουμε υπόψη μας ε, και να μην κάνουμε τίποτα. Επίσης, η συνθήκη για την εμπορία όπλων βάζει ορισμένα όρια σε σχέση με το τι επιτρέπεται και τι όχι. Θα πρέπει να δούμε γεωπολιτικά και ανθρωπιστικά δεδομένα υπόψη μας. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα ε, που θα μπορούσαν να αναφερθούν. Ας περιοριστούμε στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο γιατί θα πρέπει η άμυνα να εξαιρείται ε, από τις ε, κλιματικές αλλαγές και τις προσπάθειές μας. Η διαφάνεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να, επίσης να αναφερθούν. Τέλος, ε, θα ήθελα να αναγνωρίσω την πρόοδο που έγινε στις πρώτες συναντήσεις στο άρθρο 4, για παράδειγμα, χάρη στο καλό πνεύμα του εισηγητού και όλων των σκιωδών. Ε, θα πρέπει όμως ε, να συζητήσουμε προσεκτικά τα θέματα που έχουν τεθεί εδώ και τις κατατεθήσεις τροπολογίες και να μην χρησιμοποιήσουμε την πίεση χρόνου και τις προθεσμίες προσχηματικά. Ευχαριστώ για την Άλντε, ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι άρρωστος και η φωνή μου δεν είναι πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ποιότητα της εργασίας του αλλά και την ποιότητα της συνεργασίας μας που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά όσον αφορά την πρώτη κοινή μας συνάντηση. Θα ήθελα να πω ότι όπως το είπε άλλωστε και ο Πρόεδρος, πρόκειται για ένα φάκελο ιδιαίτερα σημαντικό που ανοίγει ή ε, ξανανοίγει μια νέα εποχή όσον αφορά την πολιτική άμυνας στην Ευρώπη και που είναι διάδοχη κατάσταση ενός πιλωτικού προγράμματος. Είναι γεγονός ότι η κυριαρχία των κρατών περνάει από την κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί σε όρους ε, και στο πεδίο της άμυνας ε, να αντιδράσει και να ανταποκριθεί ε, μόνη της στις απαιτήσει της παγκοσμιοποίησης. Το θέμα είναι εξειδικευμένο και γι' αυτό τίθενται ζητήματα όπως είναι το απόρριτο, η συνεργασία με τρίτες χώρες, θέματα ευρεσιτεχνίας, θέματα εξοδυνατότητας εξαγωγών, διανοητικής ε, ιδιοκτησίας κλπ. Βεβαίως ε, υπάρχουν προβλήματα ηθικής, δεοντολογίας, κλίματος, ε, φύλου να τεθούν και στο φάκελο αυτό. Ωστόσο δεν θα πρέπει τα σημεία αυτά να αποτελέσουν εργαλεία ελέγχου ε, σε έναν τομέα που απαιτεί ιδιαίτερα ε, προσόντα και εν πάση περιπτώσει παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Ε, ναι, είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αναφερθούν, αλλά δεν θα πρέπει ε, να αποκτήσουν υπερβολικά μεγάλες ε, διαστάσεις. Η ανάπτυξη τέτοιων πολιτικών είναι απαραίτητη, γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία σε πνεύμα συνθετικό και σε πνεύμα συμβιβαστικό. Θέλουμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις ε, οι οποίες ε, να μπορούν να αντιμετωπίσουν όσο γίνεται ευρύτερα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος από τους πρασίνους? Όχι, από την ΚΟΕ. Όχι, κανείς από την ΚΟΕ. So we've um, Από την FDD. ΕΝΕΦ. Η κυρία Λεσεβαλιέρ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη, γιατί όπως γνωρίζετε, εγώ έχω προτείνει την απόρριψη της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τροπολογία μου. Όπως έχω πει, είναι η βιομηχανική πτυχή αυτή η πρόταση μιας αθέμητης ε, ευρωπαϊκής άμυνας, δηλαδή μια αλληλεξάρτηση μεταξύ της βιομηχανίας και των ε, ενόπλων διάμενμών μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα ε, το οποίο θέτει, δημιουργεί, θέτει ε, πρόβλημα ως προς τα προνόμια των κρατών ε, μελών στην ίδια την άμυνά τους. Μου φαίνεται λογικό να υπάρχει μια ευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία ναι μεν θα μπορεί να ε, αναλάβει την άμυνα για την Ευρώπη, όχι όμως ε, να γίνει εξωτερική ανάθεση σε ε, άλλες ε, χώρες, τρίτες. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε, για παράδειγμα, το Ισραήλ μια τέτοια χώρα. Δεν νομίζω ότι πρέπει πρωτότυπα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα χρηματοδοτήσουμε. Δεν θα πρέπει να ισχύει υπεργολαβία σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο αν η τεχνολογία είναι απαραίτητη και εκ των για ε, το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω τις διάφορες τροπολογίες που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, ε, όπως για παράδειγμα εξαγωγή των ε, τεχνολογιών που προέρχονται από το πρόγραμμα, χωρίς την έγκριση της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Η κυρία Γκρίφιν θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να ασχοληθούμε ως Ευρώπη με την άμυνα και χαίρομαι ιδιαίτερα που το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει ε, το EDIDP και ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε ε, τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Πρέπει να εξισορροπήσουμε ε, την χρηματοδότηση με την καλύτερη διαχείριση γιατί δυστυχώς υπάρχουν διάφορα σκάνδαλα ε, δοροδοκίας ε, και κακοδιαχείρισης με στις δημόσιες, ε, στις δημόσιες προμήθειες ε, πρέπει ε, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ε, ενδεχομένως ένας τρόπος είναι να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες. Επίσης η αλυσίδα ανεφοδιασμού πρέπει να μην δίνει πάντοτε τη δυνατότητα σε τρίτες χώρες να είναι υπεργολάβη. Πρέπει η όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι το Ταμείο μπορεί να βοηθήσει όσον αφορά στο, στο κλίμα ε, επειδή μειώνει το οικολογικό αποτύπωμα των ενόπλων δυνάμεων όμως δεν υπάρχει καμία αναφορά ε, μεταγενέστερα στο κείμενο πέρα από την πρώτη αναφορά Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν ε, τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του Ευχαριστώ πολύ Κυρία Γκρίφιν, θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο? Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λοιπόν, από τη Γενική Διεύθυνση Γκρό. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ε, εισηγητή για την έκθεση ε, που μας παρουσίασε, που υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποιες παρατηρήσεις θα θέλαμε να κάνουμε. Ε, επειδή ο στόχος είναι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής άμενας, ε, εμείς εκτιμούμε ότι πρέπει να στοχεύσουμε ε, και να προωθήσουμε κυρίως ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως έγινε και για το EDIDP. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιο είδους συνεργασίας με επιχειρήσεις συγκεκριμένες τρίτων χωρών, αλλά αυτό αποτελεί μια εξαίρεση και θα ήταν πλαισιωμένες ε, με τον τρόπο που ε, ανέφερε, αναφέραμε και ε, στην περίπτωση του προγράμματος EDIDP. Δεν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά να υπάρξει συνεργασία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συνεργάζονται βραχυπρόθεσμα. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην υποστηρίξει κανείς τέτοιου είδους προγράμματα. Επίσης, ε, στην προπαρασκευαστική διατύπωση βαζιστήκαμε, αλλά όπως ε, θα διαπιστώσατε, προτείνουμε και κάποια εξέλιξη της ε, διατύπωσης να δούμε δηλαδή το κατά πόσο αυτό το 5% είναι σωστό ή αν είναι ένας πάρα πολύ αυστηρός κανόνας ε, μας ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ αυτή ε, η αρχή της ε, ε, διακοπής σε περίπτωση που χρειαστεί. Κάτι ακόμη πολύ σημαντικό παρατήρηση για τον δεοντολογικό έλεγχο, γι' αυτό προβλέψαμε, όπως είχε γίνει και στο EDIDP, Μόνο τα ερευνητικά προγράμματα που είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα είναι επιλέξιμα και επίσης ε, προβλέψαμε έναν έλεγχο της εφαρμογής ε, της έρευνας ε, και ελπίζουμε ότι έτσι ανταποκρινόμαστε στην ανησυχία δεοντολογικής φύσεως διατηρώντας μια ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και αν θέλετε ευχαρίστως να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να βελτιώσουμε τη σχετική διατύπωση. Και ένα τελευταίο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, εφόσον είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα, δεν είναι ένα διακυβερνητικό πρόγραμμα, δεν αυτονόητο αυτό. Ε, Κοίτα, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα έχει έναν σημαντικό ρόλο αλλά πρέπει να υπάρχει έλεγχο σε κοινοτικό επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σιγητά, κύριε Κρασνοντέμσκι, μπορείτε να συνοψίσετε τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι παρατηρήσεις. Ναι, Πρέπει να επεξεργαστούμε τη διατύπωση. Θα επεξεργαστούμε τις ε, τροπολογίες σε συμβιβαστικές. Υπάρχουν όμως ιδιαιτερότητες ε, στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Πρέπει να το λάβουμε αυτόν υπόψη και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι πελάτες είναι τα κράτη-μέλη. Και συνεπώς Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εντό του οποίου πρέπει να κινηθούμε. Είπατε ότι είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα εκπρόσωπε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμω τα κράτη-μέλη και οι ένοπλε δυνάμει των κρατών μελών θα αγοράσουν αυτό το, αυτά τα προϊόντα και συνεπώς η διακυβερνητική διάσταση είναι και αυτή αρκετά παρούσα. Πρόκειται για ένα ζήτημα συνδυασμού της καινοτομίας με την ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων. Συνεπώς πρέπει να ληφθούν υπόψη δεοντολογικά ζητήματα, το ζήτημα των κριτηρίων ε, συμμετοχής. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι δεν πρόκειται για χρηματοδότηση μη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το θέμα είναι πώς ορίζεται το ευρωπαϊκός. Και θα χρειαστεί να δώσουμε αυτόν τον ορισμό ώστε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα να αντικατοπτρίζονται. Επίσης υπάρχει και διαφορε... είναι και διαφορετική κατάσταση της άμυνας στα διάφορα κράτη-μέλη Το θέμα της προστιθέμενης αξίας είναι επίσης πολύ σημαντικό αλλά δεν μπορούμε από τώρα να πούμε ποια είναι τα αποτελέσματα του EDIDP. Ελπίζω όμως ότι με τα αποτελέσματα αυτά, ε, με τα αποτελέσματα αυτά θα μας χαροποιήσουν στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 21 Νοεμβρίου. Τώρα Πάμε στο 23 για τον ΕΝΙΖΑ, τον κανονισμό τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφορίας. Η συγγήτριά μας είναι η Αγγέλικα Νίμπλερ. η κυβερνοασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Έχει ε, αρχίσει ε, ο τριμερής διάλογος. Η εισηγήτρια θα μας πει δύο λόγια. Να μας πείτε τη γνώμη σας, πώς πάνε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαρίστως να σας πω. Στην Επιτροπή τον Ιούλιο δόθηκε εντολή για τον τριμερή διάλογο, επιβεβαιώθηκε το Σεπτέμβριο. Από τότε είχαμε δύο άτυπες, άτυπους τριμερείς διαλόγους και ευχαριστώ τον Πρόεδρο για την προσωπική του παρουσία και που, που προείδρευσαν και που, και που ευχαριστώ που προεδρεύσατε. Ε, έχουμε για τις αρμοδιότητες τη ΕΝΙΖΑ ένα διάλογο και μετά ένα καλό σύστημα πιστοποίησης στην Ευρώπη. Τώρα προγραμματίζεται το Νοέμβριο ε, κι άλλος τριμερής διάλογος και θέλουμε στις 28 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Δυο ε, τριμερείς, ένας ακόμη και μετά κλείσιμο. Αυτά διαδικαστικά. Τώρα, επί της ουσίας, θα είμαι σχετικά σύντομη. Το πρώτο μεγάλο θέμα είναι τι αρμοδιότητες, τι καθήκοντα θα έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ΕΝΙΖΑ. Εμείς στο Κοινοβούλιο είμαστε υπέρ μόνιμης εντολής με αύξηση του προσωπικού και διπλασιασμό του προϋπολογισμού. Εδώ δεν έχουμε μεγάλες διαφορές με το Συμβούλιο. Θέλουμε όμως ο ΕΝΙΖΑ να είναι μάχημη λειτουργική μονάδα γιατί υπάρχουν πολλές ε, επιθέσεις στο Μονοκράι, Πέτια και αυτά είναι, έχουν διαστάσεις που ξεπερνούν το ένα κράτος μέλος μόνο, οπότε είναι ευρωπαϊκό το θέμα, χρειάζεται καλύτερο συντονισμός για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ισχυροποίηση του ΕΝΙΖΑ λοιπόν με ίδιες αρμοδιότητες, αυτό ζητάμε. Τα κράτη-μέλη βλέπουν μάλλον υποστηρικτικό το ρόλο του ΕΝΙΖΑ. Ελπίζω να βρεθεί μία λύση συμβιβαστική. Δεύτερο θέμα για τις μορφές πιστοποίησης, κυρίως ε, συζητείτε το πώς οι διάφοροι εμπλεκόμενοι, οι ενδιαφερόμενοι και η βιομηχανία θα ενταχθούν. Εμείς έχουμε, υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Τα κράτη-μέλη θέλουν ισχυρότερο ρόλο, θέλουν να δίνουν ε, οδηγίες στον ΕΝΙΖΑ σχετικά με τις εθνικές μονάδες κυβερνοασφάλειας. Εμείς είπαμε ότι αυτό πρέπει να περνάει από την Κομισιόν, αφού ο ΕΝΙΖΑ είναι ευρωπαϊκός οργανισμός και δεν είναι εντολοδόχος των κρατών μελών. Μετά μια συζήτηση για το αν χρειάζεται υποχρεωτική ε, πιστοποίηση, όταν είναι κρίσιμη η υποδομή, τότε θα πρέπει να υπάρχει ε, ε, υποχρεωτική πιστοποίηση. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα, είναι καινούργιο οπότε δεν υπάρχουν πρόοδοι εδώ και για, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο καταναλωτής στον Οργανισμό για την ασφάλεια γιατί και ο καταναλωτής παίζει μεγαλύτερο ρόλο και θέλουμε ε, στα πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει και ενημέρωση από τον ε, κατασκευαστή ή τον ε, προμηθευτή. Και εδώ υπάρχει κάποια επιφύλαξη από τα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο δεν είναι έτοιμο να ε, στηρίξει αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά δεν είναι και ξεκάθαρα κατά. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουν. Συνοπτικά λοιπόν πρέπει να πω ότι δεν τα πάμε και άσχημα. Αρχίζουν να διαφαίνονται οι διαφορές, ότι τα κράτη λένε ότι είναι βασική αρμοδιότητά μου τα κράτη-μέλη. Ε, η κυβερνοασφάλεια. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν και εμπειρογνωμοσύνη, έχουν και ε, know-how και πρέπει να δούμε την ευρωπαϊκή διάσταση όμως τώρα. αυτά είναι που συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ, είσαστε πολύ ξεκάθαροι. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Ο κύριος Παουλ Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ. Ο ΕΝΙΖΑ είναι πολύ σημαντικός για την ψηφιακή εσωτερική αγορά και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη σε διεθνές επίπεδο. Εμείς θέλουμε να έχω, υπάρχει εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο και με ενδιαφέρει ο Ενίζα είναι καλά εξοπλισμένος και λειτουργικός και αποτελεσματικός. Ε, επίσης ε, οριζόντια συνδέεται με τον Μπέρεκ για την ψηφιακή αγορά και τους ρυθμιστικούς φορείς. Είναι σημαντικό να υπάρχει διασύνδεση και όταν ε, στο ηλεκτρική ενέργεια θέλουμε μια λειτουργική αγορά τότε χρειάζεται συνεργασία και με Μπέρ και Ενίζα. Διότι το δίκτυο λειτουργεί και μπορεί να είναι βέλτιστο μόνο αν έχει ψηφιακή διασύνδεση. Σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθεί ο ΕΝΙΖΑ και ε, προτεραιότητα για μας είναι ο ρόλος του ε, με τα ε, υφιστάμενα δίκτυα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Είσαστε σαφείς. Αγγέλικα, θέλεις να πεις κάτι? Όχι. Καλώς. Σας θυμίζω ότι αυτό ήταν το σημείο 23 στην ημερήσια διάταξή μας. Τώρα ξαναγυρίζουμε στο σημείο 17. Θέσπιση προγράμματος ε, για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Ο εισηγητής μας ε, είναι και η συγγήτρια, είναι η αντιπρόεδρος κυρία Πατρίσια Τόγια. Το πρόγραμμα, το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, συνδυάζει τέσσερα υφιστάμενα προγράμματα. Το ένα είναι το κόσμε. και βάσει του άρθρου 54 του κανονισμού έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για οποιοδήποτε ε, θέμα αφορά το κόσμε. Και ε, έχουμε και επιμερισμένη η ε, κοινή αρμοδιότητα με τις επιτροπές ΙΜΚΟ, ΕΝΒΙ, ΕΚΟΝ για οριζόντια ε, κομμάτια της έκθεσης. Ε, έχουμε λοιπόν για το κόσμο αποκλειστική και κοινή αρμοδιότητα στα άλλα θέματα με τις άλλες επιτροπές. Κυρία Πατρίσια Τρόγια, Τόγια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι έχουμε εδώ αρμοδιότητες μοιρασμένε με άλλες ε, ε, επιτροπές και ο Πρόεδρος ε, αγωνίστηκε, έδωσε μάχη έτσι ώστε στο Προεδρείο να, στη το των Προέδρων συγκεκριμένα, να μπορέσει να κρατήσει για τη δικιά μας Επιτροπή ακέραιο το ε, ε, πλαίσιο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε Μπούζεκ. Όσον αφορά τώρα το δικό μας τμήμα, εδώ αναφερόμαστε ε, στον επαναπροσδιορισμό του προγράμματος COSME. Πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι το πρόγραμμα αυτό λειτουργήσε καλά, ωστόσο δυστυχώς είχε λίγες, λίγους πόρους στην διάθεσή του. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε μια εικόνα της Ευρώπης αρκετά κοντά ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εν πάση περιπτώσει θετική εικόνα. Στην πόλη μου και στην ε, ε, περιφέρειά μου ήρθα σε επαφή με πολίτες, φαντάζομαι και άλλοι έκαναν το ίδιο και σε γενικές γραμμές είναι θετικό το πρόσημο το οποίο βάζουν οι πολίτες σε αυτήν την διαδικασία. Είναι γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές ακόμα περισσότερο, δυσκολεύονται πάρα πολύ να να περάσουν στην επόμενη φάση και μετά από την οικονομική χρηματοπιστική κρίση από τη μία ε, και από την κρίση που προκύπτει από την μεγάλη παγκοσμιοποίηση ε, απέναντι σε αυτές τις κρίσεις λέω οι αυτές οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Ε, είναι γεγονός λοιπόν ότι η σημασία του κόσμου και για το μέλλον είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αφορά κοινοτική ενωσιακή υποστήρεξη ε, σε, ε, στην ε, καινοτομία, τεχνολογική καινοτομία, τεχνολογική, οργανωτική καινοτομία για αυτούς ας πούμε που θέλουν να κάνουν πέρα από τα προγράμματα τεχνολογικής προσαρμογής και προγράμματα κατάρτισης αυτές τις νέες τεχνολογίες, χρειάζονται νέα, νέες δεξιότητες, νέες οργανωτικές δομές ε, και επομένως πέρα και βεβαίως ε, πέρα από όλα αυτά υπάρχει και το θέμα της πρόσβασης στην τραπεζική ε, πίστη έτσι ώστε οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις να περάσουν στο επόμενο στάδιο και το ίδιο ισχύει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια λυσίδα αξιών σημαντική σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει να σας πω ότι ε, ε, λυπούμε λίγο, απογοητεύομαι λίγο, το κόσμο έχει πνιγεί κατά κάποιο τρόπο ε, πιεζόμενο από όλα τα άλλα στοιχεία στρατηγικής κλπ. Η ορατότητά του είναι μικρή, θα έπρεπε να έχει μία ξεχωριστή αναφορά το πρόγραμμα αυτό έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ακριβώς περί τίνος πρόκειται και να ανεβεί λίγο και το brand name πούμε ε, του κόσμου. Θα πρέπει να ενισχυθεί λοιπόν το σήμα και να ενισχυθεί και ο προϋπολογισμός. Είναι παράλογο η Κομισιόν να μειώνει τον ε, προϋπολογισμό ε, ενός προγράμματος που έχει ήδη λειτουργήσει. Το είπε και ο, ο ίδιος ε, ο, ο Επίτροπος Τιγκέρ ότι πρέπει να υποστηριχθούν οι καλές εμπειρίες. Μπορούμε επίσης να αναπτύξουμε περισσότερο το είδος των δράσεων που θα πρέπει να λάβουν χώρα. Είπα και προηγουμένως κατάρτιση για νέα προσόντα και δεξιότητες, κατάρτιση για την επιχειρηματική κουλτούρα για την επιχειρηματικότητα. Μπορούμε επίσης να ενισχύσουμε και κάποια άλλα στοιχεία του προγράμματος αυτού. Για παράδειγμα, το ευρωπαϊκό δίκτυο των, ή μάλλον το δίκτυο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, ε, αφού έχει λειτουργήσει καλά μέχρι τώρα, να δει τον ρόλο του ενισχυμένο. Η Κομισιόν ίσως θα πρέπει να μελετήσει ε, το δίκτυο αυτό και να δει πού μπορεί να το βελτιώσει. Γιατί ε, αυτό το European Enterprise Network μπορεί να έχει κάποια στοιχεία τα οποία λειτουργούν καλά, ε, που βοηθούν εταιρείε και τα λοιπά, επιχειρήσει και κάποια, σε κάποιε άλλε χώρε να μην λειτουργεί πάρα πολύ καλά γιατί οι νομικέ δομέ είναι διαφορετικέ. Εγώ και το προτείνω μέσω τροπολογία. θα ήθελα να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Η κοινωνική οικονομία αγορά μας αναφέρεται ε, ε, ε, στα χαρτιά αλλά λίγα κάνει η Ευρώπη για αυτό το θέμα. Μιλάμε εδώ για επιχειρήσεις ε, οι οποίες δεν ε, ε, απέλησαν προσωπικό, έχουν δείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, μεγαλύτερη αντοχή γιατί λειτουργούν επιτόπου και έχουν καλύτερη επικοινωνία, καλύτερη, μεγαλύτερη δύναμη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα έλεγα να έχουν πρόσβαση στον κόσμο και αυτού του είδους οι επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ε, α, και κάτι τελευταίο. Εδώ το έρασμος ε, και το κόσμο είναι γνωστό ε, παντού. Και γιατί λοιπόν θα πρέπει να βγάλουμε το όνομα αυτό από μια καινοτομία η οποία έχει λειτουργήσει καλά και όλοι ξέρουν το όνομά της. Υπάρχουν προγράμματα όπως το Horizon, το Invest EU και το COSME τα οποία πρέπει να προωθηθούν. Ευχαριστώ. Σας Ευχαριστώ. Θα έχετε και την να, δυνατότητα. Θα πω δύο λόγια. Ε, θα, πείτε δύο λόγια μετά. Η τώρα. Ο κύριος Ρούμπικ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Τόγια θερμά. Ε, γιατί είναι στην καρδιά του θέματος. Εμείς ε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε πάνω στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα TIP είχε αναπτυχθεί παλιότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήταν πρόγραμμα ανταγωνισμού και καινοτομία. Στην τελευταία Αυστριακή Προεδρία ε, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις και το κόσμο αισιοδοξούμε ότι ε, με την ίδια ζωντάνια θα γίνουν και διαπραγματεύσεις στην ε, ε, επόμενη μας προεδρία. Η ΜΜΕ καλύπτουν το 50% του ΑΕΠ και απασχολούν τα δύο τρίτα του εργατικού δυναμικού. Και η αύξηση των εργαζομένων είναι μεγαλύτερη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι όμιλοι μειών προσωπικό, οι μημια αυξάνονται και επεκτείνονται και σε προσωπικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης το 80% των φόρων το πληρώνουν οι ΜΜΕ η Amazon, αυτά που δεν πληρώνει, τα πληρώνουν 100% ε, ε, και πληρώνουν πλήρως τους φόρους οι μικρές επιχειρήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, ανακουφιστούν και οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπιστούν με δικαιότερο τρόπο. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές. Από τη μια πλευρά έχουμε εισηγμένες ε, εταιρείε ε, που μεγιστοποιούν τα κέρδη και αντιμετωπίζουν πιέσεις σε σχέση με τους μετόχους και έχουμε και τις οικογενειακές επιχειρήσεις όπου πρόκειται για περισσότερες γενναίες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα μέλη των επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση πρέπει να είναι στο επίκεντρο και η σταθερότητα της επιχείρησης. Γι' αυτό είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό ε, Δίκτυο να επεκταθεί και στα, νεό, στα πιο καινούργια κράτη-μέλη. Ε, υπάρχει μια μελέτη για τα νέα κράτη-μέλη και γιατί οι δαπάνες για την έρευνα και άλλα κονδύλια από τα ταμεία ε, δεν αξιοποιούνται γιατί δεν υπάρχει η απαραίτητη οικοδόμηση ικανοτήτων. Εκεί χρειάζεται να επενδύσουν. Είναι δύσκολο να κατατεθούν τα αιτήματα και να ε, τύχουν επεξεργασίας. Εμείς ε, θέλουμε αυτό το επιχειρηματικό δίκτυο να παρέμβει και να λύσει παρόμοια προβλήματα, κυρίως στα καινούργια κράτη-μέλη. Ε, έχουμε τα νέα ταμεία, το ΕΦΣΙ για στρατηγικές επενδύσεις ή ταμεία που δίνουν μεγάλα δάνεια. Πρέπει να φροντίσουμε το κόσμο να μπορεί να συμμετέχει σε όλα αυτά. Ε, όπως παλιότερα ε, συνέβαινε με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν ιδιαίτερα στην έρευνα. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αναλάβουν το ρόλο τους. Και πιστεύω ότι ένα εράσμους για νέους επιχειρηματίες είναι ένα ιδιαίτερα ε, σημαντικό πρόγραμμα. Καλό είναι να επεκταθεί στα πλαίσια των διεθνών ανταλλαγών. Και εγώ είμαι υπέρ. Ευχαριστώ, διακόπτη ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μπασίρ για την ομάδα ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ ε, την εισηγήτρια. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η πρόταση για ε, τη ε, βιομηχανία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μένουμε επικοδομητικές συζητήσεις μαζί της και τους υπόλοιπους σκηχιώδεις εισηγητές. Το σχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει σημαντικές προτάσεις. Βέβαια, το κόσμο για μας είναι μία προτεραιότητα για την ομάδα μου αλλά και για ολόκληρη την Επιτροπή μας. Έχει γίνει αποδεκτό πολύ καλά από τον κλάδο και ελπίζουμε να υπάρξουν αποτελέσματα ε, στο επόμενο Ε, βελτιώνει το σχέδιο γνωμοδότησης ε, την πρόταση για παράδειγμα ε, τις οι κοινωνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και οι προτάσεις της επιτρέπουν ε, να μην υπάρχει αυτή η πόλωση μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών ε, επιχειρήσεων θα μπορούσαμε με τη συνεργασία τους να καταλήξουμε σε οικονομίες κλίμακας. Ε, για παράδειγμα, η δειγματοποίηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, θέμα για την ενίσχυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Όσον αφορά τις ε, ανεπάρκειες της αγοράς, καταλαβαίνουμε την πρόθεση, αλλά δεν υπάρχει επαρκής ορισμός για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα προτιμούσαμε να παραμείνει εκτός αυτό το κομμάτι. Επίσης, όσον αφορά την προώθηση της απασχόλησης, ε, ε, και ε, επειδή μιλούσαμε για πολύ χρήσιμες ιδέες, δεν τις βλέπουμε, δεν είναι πολύ σαφείς και δεν βλέπουμε πώς μπορούν αυτοί οι στόχοι να επιτευχθούν μπορούμε να υποστηρίξουμε, με την ενίσχυση, να υποστηρίξουμε την ενίσχυση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα προγράμματα παρακολούθησης μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα, ειδικότερα για ομί... ομίλους, που... για ομάδες που δείχνουν μικρότερη τάση προς την επιχειρηματικότητα. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να έχει μια διεθνή διάσταση αυτό το πρόγραμμα, ενίσχυση δηλαδή ε, βιομηχανική και ρυθμιστική συνεργασία με τρίτες χώρες. Αυτά τα μη δασμολογικά εμπόδια αυξάνουν ε, τα προβλήματα ενώ ε, πολύ μεγάλες ας πούμε πολύ μεγάλα, μεγάλες δυνάμεις δεν αναγνωρίζουν η μία την άλλη. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχουν ε, κάποια υποστηρικτικά μέτρα για να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε τις ε, συνέργειες ε, με τα άλλα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που άργησα ε, και προς την εισηγήτρια αυτής της ε, γνωμοδότησης που εξετάζουμε αλλά και από τους προηγούμενους εισηγητές. Δυστυχώς είχα κάποια θέματα στην Επιτροπή Μεταφορών που συνέπιπταν χρονικά με τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι επικροτώ την πρόταση. Πιστεύω ότι η ολοκλήρωση είναι το σωστό, η σωστή κατεύθυνση. Απλώς... δεν ξέρω αν υπάρχει επαρκής εστίαση στις προτεραιότητες και παράλληλα στη μείωση του διοικητικού φόρτου. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσω, είναι κάτι το οποίο ε, παραμένει προς ε, αποσαφήνιση. Κρίμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας υπόψη ότι υπάρχει φιλοδοξία στο Συμβούλιο μεταξύ των ε, πολλών κρατών μέλων, ήταν κάπως μετριοπαθής όσον αφορά του ε, δεδομένου του πεπέδου του προϋπολογισμού. Ε, δεν νομίζω ότι αντανακλά τη σημασία του προγράμματος αυτού ε, δεδομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών του και των διαφόρων συνιστοσών του. Ε, όσον αφορά την ε, έκθεση της κυρίας Τόγια, θα έλεγα ότι είναι πολύ καλή. μπορώ να συμφωνήσω με την ε, μεγάλη πλειοψηφία των προτάσεών της. Ε, χαίρομαι που ε, αναφέρθηκε στο θέμα του προπολογισμού, επειδή το ανέφερα και εγώ και ελπίζω να υπάρξει συμβιβασμό στο μέλλον όσον αφορά την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης, πράγματι συμφωνώ απολύτως με το συλλογισμό της που μας τον εξήγησε όσον αφορά τώρα την τοπική δημόσια επιχείρηση, ορισμός που έχουμε εδώ έχω μια μικρή δυσκολία. Είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψουμε περαιτέρω. Οι ιδιωτικές εταιρείες ε, επιφορτίζονται με το ε, φόρτο αυτό και θεωρώ ότι υπάρχει ένα, έχουν ένα μειονέκτημα ε, σε σχέση με τις δημόσιες και ίσως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το λύσουμε αυτό. Επίσης εκτιμώ την προσπάθεια της εισηγήτριας ε, στο άρθρο 3 ε, και το στόχο 8 ε, να είναι πιο επιλέξιμα τα συγκεκριμένα προγράμματα. Είμαστε υπέρ σε γενικές γραμμές της γνωμοδότησης της ηγήτριας και με χαρά θα περιμένουμε τις συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, εκ μέρους των Πρασίνων, κυρία Μέτς. Ευχαριστώ συνάδελφοι, κυρία εισηγήτρια, ευχαριστώ την κυρία Τόγια για την εξαιρετική δουλειά στο σχέδιο γνωμοδότησης. Τονίζω ότι χθε το IPCC θέσπισε ειδική έκθεση που είναι ακρογωνιαίος λίθος για τη Συμφωνία των Παρισίων. Μέχρι το τέλος του αιώνα μπορούμε να μειώσουμε κατά 1,5 βαθμό τη θερμοκρασία, αλλά αυτό είναι καλό. Αλλά το κακό είναι ότι οι πολιτικές μας δεν ε, είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να το κάνουν. Θα πρέπει να συμβάλλουμε στη μείωση της χρήσης άνθρακα και στο στόχο τουλάχιστον 30% δαπάνες ε, για το κλίμα στο πολιετές δημοσιονομικό. Συμφωνώ με κάποιες ε, ε, ε, τροπολογίες σας, άκουση του προϋπολογισμού για τις ΜΜΕ ή μονοθυριδικές υπηρεσίες για την πρόσβαση. Όμως τρία πράγματα θα τονίσω που μου έκαναν εντύπωση στην πρόταση της Κομισιόν. Πρώτον, η βιωσιμότητα. Στην πρόταση της Κομισιόν ε, αναφέρεται η έννοια της βιωσιμότητας και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες που έχουν γίνει ε, έχουν, ε, έχουν τύχει επεξεργασία. Στο κόσμε επίσης ε, γίνεται αναφορά όπως και σε πολλούς δείκτες βιωσιμότητας. Αυτοί όμως δεν υπάρχουν στην πρόταση της Κομισιόν τώρα. Η βιωσιμότητα πάει χέρι με χέρι με την ανταγωνιστικότητα και ε, δίνει μεγάλες ευκαιρίες στις, ε, κυρίως στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς. Θα καταθέσω με που θα παρουσιάζουν πιο συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας, όπως και δείκτες. Δεύτερον, η παρακολούθηση και οι αναφορές, οι εκθέσεις ε, είναι πολύ σημαντικές. τώρα είναι αφήσεις ό,τι αφορά το κόσμο. Καταλαβαίνω ότι όταν μιλάμε για την προστασία καταναλωτών, την ανταγωνιστικότητα, τις στατιστικές, όλα μαζί, συνολικά είναι δύσκολο να τεθούν προϋποθέσεις για παρακολούθηση και ε, αναφορές. Ε, πρέπει όμως να, για χάρη των παραληπτών να ξέρουμε σε τακτή βάση τι συμβαίνει για να εντοπίζουμε ελλείψεις αλλά και τα θετικά στοιχεία του προγράμματος. Ε, κάποιες προϋποθέσεις πρέπει να οριστούν λοιπόν για αυτό το λόγο και θα το εξετάσω πιο συγκεκριμένα το θέμα. Τέλος, ε, οι ειδικέ ανάγκες των ΜΜΕ. Όπως ε, αναφέρει σωστά η κυρία Τόγια στο κόσμο ε, ήταν εύληπτη η γλώσσα για τις ε, ομάδες στόχο που θα μπορούσαν να χρειάζονται εκπαίδευση ή μια επιχειρηματική κουλτούρα και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις ΜΜΕ, μείωση του διοικητικού φόρτου κλπ. Πιο αργά ε, ε, να μιλάτε, λέει ο πρόεδρος. Πέρασε και ο χρόνος σας. Τελειώνω. Οι μονοθυριδικές υπηρεσίες θα ήταν καλές. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια και περιμένω τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Συγγνώμη, αλλά δεν πρόσεξα το χρόνο. Ζητώ συγγνώμη και από τους διερμηνείς γιατί ίσως καθυστέρησα να σας επισημάνω ότι δεν πρέπει να μιλάτε με τέτοια ταχύτητα. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε λέει η κυρία Μέτς. Ο κύριος Κοχλίτσεκ θα, αντικα... Ε, θα αντικαταστήσετε την κυρία Παλώμα Λόπες Μπερμέχο που είναι σκιώδης. Ναι, ναι, ε, δεν θα μπορέσω να σταθώ στο ύψος της, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και ό,τι καταφέρω. Οι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, όπως λέει άλλωστε και η ίδια η εισηγήτρια, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Στην ε, Τσεχία έχουμε εμπειρία εντός εισαγωγικών ε, όσον αφορά το γεγονός ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις λίγο συμβάλλουν στον κρατικό κορβανά και τον κρατικό προϋπολογισμό γιατί συχνά έχουν προγράμματα φοροαποφυγής κλπ. Ενώ αυτές οι μικρές επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν να το κάνουν και επομένως πληρώνουν ε, φόρους. Επίσης πολύ συχνά έχουμε εταιρείες ε, οι οποίες ενώ ενώ είναι τσεχικές και δρούν στην Τσεχία, έχουν δημιουργήσει έδρες ε, και ε, εταιρείε ε, εκτός της Τσεχίας. Αυτό εννοώ κιόλας και φορά αποφυγή. Ε, οπωσδήποτε ε, είναι πολύ θετικό αυτό που ζητάει η συγγήτρια να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικού προσήμου επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν ε, ε, τις ε, κοινότητες ε, και στους δήμους. Είναι πολύ σημαντικό ε, οι διοικητικέ διαδικασίες να είναι απλές. Αυτή η ενιαία θηρίδα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική και να πω στην εκπρόσωπο των Πρασίνων που μίλησε πριν από εμά ότι εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσουμε λίγο περισσότερο το πράσινο στοιχείο. Υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις ή μικρή ε, παραγωγή ανανεώσιμων ε, ε, ειδών ενέργειας που δεν έχουν εξαιρετική κατάσταση, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Άρα καλά να κάνουμε κάτι για τους ε, και για αυτούς τους μικρούς προμηθευτές ε, ενέργειας, να τους βοηθήσουμε όσον αφορά ας πούμε τα διοικητικά στάδια και τα λοιπά και όχι μόνο τους εμπόρους και ε, αυτούς του επιχειρηματίες. Ευχαριστώ και θα συνεχιστεί καλά η συνεργασία με την κυρία Τόια. Η κυρία Αμάτο. Από την FDD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γνωρίζουμε το όλοι ότι ε, η παγκοσμιοποίηση δημιούργησε πολλά προβλήματα, προκάλεσε πολλά προβλήματα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ε, δίνοντας ε, προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο και σε επίπεδο αποσχόλησης που γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχει ανάγκη εναρμόνισης ε, του ε, θεσμικού πλαισίου ε, και οπωσδήποτε η πρόσβαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και η προστασία των καταναλωτών είναι θέματα πολύ σημαντικά. Χρειάζεται μία πιο αποφασιστική καμπή έτσι ώστε να βοηθηθούν κυρίως οι μικρές, μεσές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επίσης η συλλογή των στατιστικών στοιχείων ακόμα και μη ομαδοποιημένων ε, να χρησιμοποιηθούν ε, έτσι, έτσι ώστε να υπάρχει οικοβιωσιμότητα και για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία, μέχρι το 2050 σε μια οικονομία ε, η οποία θα έχει απελευθερωθεί από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης όσον αφορά το Invest EU ε, θα έπρεπε να απαγορευθούν όλες οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλο, υπερβολικά μεγάλο κίνδυνο. Ε, και θεωρούμε ότι θα πρέπει ε, όλες ε, οι δυνατότητες οι οποίες δίνονται στις υπηρεσίες και στους επιχειρηματίες να έχουν περάσει πρώτα από κόσκινο και να, είναι, να μην παρουσιάζουν επικινδυνότητα. Κάτι άλλο, ένα άλλο στοιχείο το οποίο θεωρούμε σημαντικό για την λήψη πολιτικών αποφάσεων. Εάν εκτός από το ΑΕΠ βρούμε το θάρρος να βάλουμε και δείκτες που θα μετρούν την κοινωνική κοινωνική κατάσταση ε, και την ε, οικολογική βιωσιμότητα εάν μπορέσουμε να, συνυπο, να συνμετρήσουμε ε, ε, και στοιχεία όπως είναι ας πούμε η μόλυνση κλπ. Πιστεύουμε ότι και στους πολίτες μας και στις επιχειρήσεις μας ε, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον. Κατά την έννοια των λεγόμενων μου θα υποβάλουμε και τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή κυρία, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Σράιμπερ. Έχει το λόγο. Παναγιά υπεύθυνοι για το κόσμο πρέπει να πω ότι πάντοτε μας υποστήριζε η Επιτροπή σας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Βάσει της αξιολόγησης του κόσμε που ήταν πολύ θετική γενικά, ε, καταρτήσαμε αυτή την πρόταση ε, για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς που είναι σημαντικό πυλώνας για τις ΜΜΕ. Μπορέσαμε να χτίσουμε πάνω στο, ε, στην καλή δουλειά που έγινε κατά το παρελθόν και να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις. Ε, σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι η θέση των ΜΜΕ ε, είναι γνωστή. Θέλουμε πολιτικές ανάπτυξης ε, για τα χρηματοδοτικά μέσα ε, θα φροντίσουμε να υπάρχουν μεγάλες συνέργειες και να συνεχίσει να υπάρχει η υποστήριξη τόσο αποτελεσματική όσο και στο παρελθόν. Ευχαριστώ για τις πολλές προτάσεις για το Enterprise Europe δίκτυο. Εδώ έχουμε μια συνέχεια της στήριξης της καινοτομίας και ο κύριος Ρούμπικ ανέφερε κάποια θέματα βελτίωσης και εσείς ε, επίσης. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπου η υποστήριξη λειτουργεί καλύτερα από ό,τι αλλού, αλλά η στήριξη είναι η ναυαρχίδα και θα οικοδομήσουμε πάνω στις εργασίες που έχουν ήδη γίνει. Είμαστε ανοιχτοί στις νέες προκλήσεις και έχουμε και ειδική ομάδα εργασίας για το πώς μπορεί να ωφεληθούν από τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών ή ΜΜΕ. Όλα αυτά θα μπορούν να γίνουν χάρη στο Enterprise Europe Network ε, και την καλή χρηματοδότηση. Χρησιμότητα αναφορά στην κοινωνική οικονομία είπατε ότι χρειάζεται, ευχαρίστως να το κάνουμε. Το μόνο είναι ότι θα πρέπει να γίνει αναφορά στην κοινωνική οικονομία και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, γιατί υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις εκεί για το πρόγραμμα Εράσμους για τους επιχειρηματίες και εδώ ευχαριστούμε πολύ για την υστήριξη που μας προσφέρει η Επιτροπή σας. Πρόκειται για ένα παράδειγμα προγράμματος που είναι χαμηλών τόνων αλλά ε, πολύ φιλόδοξο. Θέλουμε να το συνεχίσουμε. Ε, το, το, το όνομα είναι πολύ γνωστό, είναι συμβουλευτικό πρόγραμμα για επιχειρηματίες και σας διαβεβαιώνω κύριε Ρούμπιχε σχετικά με το διεθνή του χαρακτήρα. Τώρα περνάμε, είμαστε στην πιλωτική φάση ε, για να διεθνοποιηθεί το πρόγραμμα και θέλουμε να συνεχίσουμε ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, για το... την κατανομή των κονδυλίων, δεν έχουμε περισσότερα ε, κονδύλια, αλλά Σίγουρα ε, χρειάζονται αναγκαίοι πόροι για το δίκτυο. Ε, δεν θα μπω σε ε, στις λεπτομέρειες των τροπολογιών. Οι δίκτες πρέπει να είναι σημαντικοί, να μην δημιουργούν γραφειοκρατικό βάρος περισσότερο. Και επίσης προσαρμόζουμε τους δίκτες στα πλαίσια του Enterprise Europe Network για να είναι ελάχιστος ο διοικητικός φόρτος και μέγιστη πληροφόρηση και θα μπούμε και σε λεπτομέρειες όταν έρθει η ώρα. Ε, θα μιλήσουμε για τις πιο τεχνικής φύσεως τροπολογίες. Γενικά πάντως ε, είμαστε ευτυχείς για την υποστήριξη που μας ε, δίνεται και είναι πολύτιμη αυτή η στήριξη για μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόγια. Γήτρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, γιατί ο καθένας ε, είπε κάτι συμπληρωματικό και υπάρχουν προτάσεις όπως του συναδέλφου Ρούμπιχ και άλλων που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ε, θα μελετήσουμε βεβαίως ε, εν λεπτομερία όλα τα στοιχεία και όλα αυτά που είπαν και άλλοι συνάδελφοι πολύ σημαντικά. Ε, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν και οι ε, ε, εταιρείε οι οποίες μπορεί να έχουν ένα κοινό προφίλ, οι οποίες μπορεί να είναι όντως σε τοπικό, κοινοτικό επίπεδο, σε επίπεδο Δήμου δηλαδή και περιφέρειας. Συμφωνώ επίσης ε, και όσον αφορά τα θέματα της βιωσιμότητας ε, που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Νομίζω ότι άλλωστε κοινή ε, κατεύθυνση ακολούθησαν όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις και εγώ μπορώ να τα συμμεριστώ όλα. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην ενδυνάμωση του, της χρηματοδότησης. Θα πρέπει να σκεφτούμε ακριβώς τις υπηρεσίες που μπορούμε να δώσουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αυξήσουμε δηλαδή τις δυνατότητες Ωστόσο, πολλές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες ε, θα ήθελαν να συμμετάσχουν αλλά δεν υπήρχαν ε, σχόλια. Δυστυχώ, ε, η ομίλητρια μιλάει πολύ μακριά από το μικρόφωνο, οι διερμηνείς δυσκολεύονται πάρα πολύ να την ακούσουν. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια σοβαρή, σωστή απάντηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και να μελετήσουμε τον λόγο για τον οποίο ε, υπάρχει τόσο χαμηλό ε, ποσοστό επιτυχίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε όλοι ένα κοινό πλαίσιο, κοινό πνεύμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ε, ε, σκιώδεις ε, για την εργασία τους και θα ακούσω τις προτάσεις τους. 15 Οκτωβρίου η υποβολή των τροπολογιών, 5 Νοεμβρίου η μελέτη εξέταση μάλλον των τροπολογιών, πρώτη ψηφοφορία στην Επιτροπή 21 Νοεμβρίου και στην αρμόδια καθήλια Επιτροπή ΙΜΚΟ 21 Νοεμβρίου του 2019. Πάει λοιπόν και το σημείο 17 της ημερησίας διατάξεως και φτάνουμε στο σημείο 18 άσερ παρουσίαση λοιπόν η οποία θα γίνει από τον Αλμπέρτο Ποτότσνικ, ο οποίος είναι διευθυντής ε, του Άσερ. Αγαπητέ κύριε Διευθυντά, να σας ζητήσω να έρθετε κοντά μας. Κύριε Ποτότσνικ, διευθυντή, διευθυντά του Acer, στις 15 Σεπτεμβρίου θα έλεγε η θητεία του, αλλά ε, εν εκτελεί χρέη ε, διευθυντή για την τρέχουσα περίοδο. Το τρίτο ενεργειακό πακέτο και η παρακολούθηση της εσωτερικής ε, αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου. Αυτό είναι το καθήκον του. Γίνεται μια αιτήσια έκθεση τεσσάρων τόμων που αφορούν ε, την, ε, τον ηλεκτρισμό, ε, τον, τις αγορές κοντρικής αερίου, δύο τόμους τις δύο τόμοι της έκθεσης ε, του 2018 για, ε, τις, ε, για το αέριο και μια προκαταρκτική για την λιανική αγορά ηλεκτρισμού έχουν ήδη δημοσιευθεί και στις 22 Οκτωβρίου οι, υπόλοιποι, οι άλλοι δύο τόμοι θα δημοσιευθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας την Επιτροπή Ήτρεν να ακούσουμε τι έχετε να μας πει κύριε Διευθυντά και να ξέρουμε ποια είναι η άποψή σας για την παρακολούθηση ε, της αγοράς, γιατί ο Acer είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα της αγοράς μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι ευρωβουλευτέ τη επιτροπή αυτής. Είναι τιμή για μένα να είμαι και πάλι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω μερικά από τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησής μας. Όπως είπε και ο πρόεδρο, φέτο και πέρυσι ασχοληθήκαμε με τον ηλεκτρισμό, τον αέριο, το αέριο, τις χοντρικέ ε, αγορέ ε, και μετά ε, την λιανική αγορά ηλεκτρισμού και την ε, προστασία των δεδομένων. Δεν θέλω να αναφερθώ στα βασικά μηνύματα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες παρακολούθησής μας. Και θα δείτε ότι κάποια από τα θετικά μηνύματα της περσινής χρονιάς επιβεβαιώνονται και κάποιες από τις προκλήσεις της αγοράς ε, επίσης. Τα καλά νέα είναι όμως ε, που, ότι κάτι που εμφανίστηκε πέρσι είναι η συμμετοχή ε, του Κοινοβουλίου ε, και ε, του Συμβουλίου στην προσπάθεια αυτή η δουλειά των εθνικών ρυθμιστών, των ενδιαφερομένων φορέων επιτέλους καρποφορούν και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ωφέλη όλης αυτής της διαδικασίας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με το θετικό μήνυμα. Οι λιανικές τιμέ, οι τιμέ λιανική πέφτουν. Ε, αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα από μόνο του, αλλά ε, πρέπει να είμαστε κάπως συγκρατημένοι ως προς αυτό, να μην υπερενθουσιαστούμε, γιατί σε κάποιο βαθμό μια αγορά κρίνεται ε, και σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις των αγορών. Ε, από πέρσι όμως επιτέλους ε, οι τιμές λιανικής ακολουθούν τις τιμές χονδρικής. Για πολλά χρόνια έχουμε δει ε, τιμές χονδρικής να πέφτουν και να αυξάνονται οι τιμές της λιανικής. Επιτέλους φέτος αυτές οι δύο τιμές, λιανικής και χονδρικής, κατά μέσο όρο ακολουθούν μια παρόμοια πορεία, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η αγορά λειτουργεί καλύτερα, γιατί τα μηνύματα για τις τιμές από ε, τις τιμές χοντρικής φτάνουν επιτέλους, ε, μετακυλίονται στον καταναλωτή. Το, το αμφισβητήσιμο κομμάτι αυτού που πληρώνουμε εμείς ως Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, μειώνεται ακόμη περισσότερο. Το αμφισβητήσιμο ε, κομμάτι είναι αυτό που καλύπτει το κόστος του αγαθού, του αερίου δηλαδή και του ηλεκτρισμού, αλλά πρέπει να πληρώσουμε και το κόστος παράδοσης της, ε, του ηλεκτρισμού ή του αερίου στα σπίτια μας, δηλαδή το κόστος του δικτύου. Και επίσης υπάρχουν μετά οι φόροι, υπάρχουν άλλα στοιχεία όπως για παράδειγμα τα τέλη που πρέπει να πληρώνουμε. Ε, αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι των όσων πληρώνουμε. Αυτό δεν είναι αξιολογική κρίση. Είναι απλώς ε, μία σκέψη που σημαίνει ότι ο χώρος για ανταγωνισμό ε, είναι ένα μικρό τμήμα, το 1 τρίτο στον ηλεκτρισμό και στο αέριο είναι κάτω από το ίμιση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν προσπαθούμε να προωθούμε τον ανταγωνισμό. Είπα ότι επιτέλους υπάρχει μια καλή και παρόμοια πορεία ε, παράλληλη των τιμών χονδρικής και ηλιανικής. Ας περάσουμε πρώτα στο αέριο. Στο αέριο βλέπουμε ότι ο κώδικας δικτύου και η καθοδήγηση που εσείς ε, εγκρίνετε τα τελευταία χρόνια έχουν αντίκτυπο στην αγορά. Ε, όλο και περισσότερη ικανότητα ε, αφορά το βραχυπρόθεσμο κομμάτι, το μακροπρόθεσμο ε, κομμάτι που είναι το μπλε, είναι το κυρίαρχο, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και το κίτρινο που είναι πάνω από αυτό και βλέπετε σιγά σιγά ότι αυτό κερδίζει έδαφος. Επίσης είναι άξιον παρατήρησης ότι υπάρχει ενδεχομένως ε, λίγο ε, μεγαλύτερη ικανότητα, αλλά ε, σε επίπεδο βραχυπρόθεσμου booking ε, βλέπουμε ότι η, η αντίδραση της αγοράς είναι καλύτερη, ε, κάτι το οποίο ε, σημαίνει ότι υπάρχει και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. Αυτό έχει βέβαια αποτέλεσμα και στην ασφάλεια ανεφοδιασμού. Εδώ βλέπετε έναν μέσο όρο που είναι ο δείκτης. Είναι η ικανότητα των διαφόρων αγορών αερίων των διαφόρων κρατών μελών να αντέξουν ε, την έξοδο ή τη μη διαθεσιμότητα μίας πηγής. Και όπως βλέπετε, κάποιες χώρες, ε, το μπλε αναφέρεται στο 2013 και το κόκκινο αναφέρεται στο 2017, που είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και όπως βλέπετε στις περισσότερες αγορές έχει βελτιωθεί η κατάσταση και τα περισσότερα κράτη είναι πάνω από το κατόφλι που είναι πιστεύουμε ε, το 110 ας πούμε ως αριθμός. Αν ε, λοιπόν ε, απομακρυνθεί η απερχόμενη πηγή να έχουμε ένα 10% περιθώριο. Αν χρειάζεσαι 110% τότε ο απερχόμενος προμηθευτής ε, ε, δεν έχει πια θέση μονοπωλιακή και όλο και περισσότερες αγορές ε, ανταποκρίνονται πλέον σε αυτήν την κατάσταση. βλέπουμε επίσης τη σύγκληση των τιμών. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο χάρτης. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη της Ευρώπης και βλέπουμε το κόστος ε, της πηγής ε, στις διάφορες ε, χώρες. Το βλέπουμε, το, το συγκρίνουμε για παράδειγμα με τους διάφορους κόμβους. Οι κίτρινες χώρες είναι οι χώρες οι οποίες είναι πολύ κοντά ως προς το ε, κοινωνικό κόστος ε, του TTF. Ε, το CL είναι 1 με 3 ευρώ και το σκούρο μπλε είναι πάνω από 3 ευρώ. Αν ξαναδείτε λοιπόν την αλλαγή μεταξύ του 2012 που είναι στα αριστερά και του 2017, βλέπετε πολύ περισσότερο κίτρινο. Ε, λοιπόν, αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερη σύγκληση τιμών. Ε, οι προμηθευτές ε, που στέλνουν σε εμά και σε πολλές ε, χώρες ε, στο περιβάλλον των χωρών της Ευρώπης μπορεί να στείλουν δηλαδή το εμπόρευμά τους, το προϊόν τους σε πολύ πιο ε, ε, ίσους όρους για να το πω διαφορετικά και επίση το κίτρινο πηγαίνει προς, από τα αριστερά προς τα δεξιά αυτό είναι περίεργο, γιατί θα έλεγε κανεί ότι οι χαμηλότερε τιμέ είναι στην, ε, σε ανατολικέ χώρε. Όχι όμω. Άρα αυτό σημαίνει ότι μια ανταγωνιστική αγορά, η προσπάθεια των ευρωπαϊκών οργάνων και άλλων ευρωπαϊκών φορέων αποδίδει. Γιατί ο ανταγωνισμό είναι αυτό που μειώνει το κόστο. Ε, αυτά είναι λοιπόν τα τρία μηνύματα τα οποία θα ήθελα να σας ε, μεταφέρω σε σχέση με το αέριο για τον ηλεκτρισμό. Το επίπεδο αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας της χρήσης των διασυνδεδεμένων δικτύων μας στο πλαίσιο ενός χρονικού ορίζοντα έχει ε, αυξηθεί και διατηρείται σε υψηλό επίπεδο 85 με 86%, δηλαδή το 85 με 86% ο αριθμός των ε, δικτύων μας χρησιμοποιείται με ε, πλήρη και αποδοτικό τρόπο. Αυτός ε, εδώ ο χάρτης μας δείχνει τις δύο μεγαλύτερες περιφερειακές αγορές ε, από το Γιβλαρτάρ μέχρι τη θάλασσα του Μπάρεν σε 19 δικαιοδοσίδες και μετά έχουμε ε, τις τέσσερις χώρες MMC Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και μετά έχουμε ε, τις ε, χώρες με ε, ροζ. Δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να επιτύχουμε πλήρη ισορροπία παρά το γεγονός ότι το UI της ενδο, των ενδοκοινοτικών κόμβων ανά ημέρα ε, ε, βελτιώνεται, οπότε ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είναι ακόμη καλύτερη εικόνα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά νέα, αλλά υπάρχουν και κάποιες προκλήσεις. Εδώ βλέπετε τις δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Η πρώτη είναι το χαμηλό επίπεδο αξιοποίησης της διασυνοριακής ικανότητας. Πιστεύουμε ότι κατά μέσο όρο στην Ευρώπη το ίμιση αυτού που θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο στην αγορά ουσιαστικά διατίθεται ε, διασυνοριακά. Αυτός εδώ χάρτης δείχνει την ε, απόδοση των διαφόρων περιφερειών ως προς τη χρήση της διασυνοριακής ε, σύνδεσης και τις διαφορές τιμών μεταξύ γειτονικών ε, ζωνών. Και βλέπετε ότι είναι λίγες οι πράσινες χώρες, άρα πολλά μπορούμε να κάνουμε ακόμη για να, δούμε, για να, μπορέσουμε, για να βελτιώσουμε το πώς χρησιμοποιούμε αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας ως προς τη διασύνδεση των δικτύων και να το μεταφέρουμε εκεί που χρειάζεται επιπλέον ικανότητα. Απ' την άλλη υπάρχει ε, η επάρκεια των πόρων. Αν δούμε ας πούμε την αξιολόγηση αυτή, βλέπουμε ότι οι χώρες που έχουν αρκετούς πόρους Βέβαια αυτό πρέπει να το δούμε και σε σχέση με τους γείτονες των χωρών αυτών, ποια είναι η κατάσταση στις ε, ε, γειτονικές χώρες και αυτή η αξιολόγηση πρέπει να γίνει σωστό, σωστά γιατί ε, υπάρχει περίπτωση να γίνει ε, διπλός υπολογισμός ή μπορεί να γίνει υπερεπένδυση ε, στην χώρα σου. Οι χώρες με κόκκινο και κίτρινο ενδεχόμενη συμμετοχή διασυνοριακών πόρων δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε άλλες χώρες λαμβάνεται υπόψη ε, βλέπετε για παράδειγμα το γκρι, το σιέλ, το σιέλ μάλλον και το σκούρο μπλε είναι αυτό, είναι οι χώρες ε, που λαμβάνουν υπόψη τις, τους διασυνοριακούς πόρους ε, με, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανότητες. εδώ βλέπουμε το πράσινο, για παράδειγμα, είναι, αυτό που βρισκόμαστε, είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις διασυνοριακές ανταλλαγές. Μετά βλέπουμε ένα κόκκινο κομμάτι που είναι η βελτίωση που προτείνουμε Προφανώς λοιπόν ε, η ολοκλήρωση των αγορών επέφερε κάποια ωφέλη. Οφέλη ε, εξακολουθούν να υπάρχουν ε, από την σύνδεση των αγορών όμως υπάρχουν, κάποιες, υπάρχουν κάποια περιθώρια ε, μεγαλύτερων ικανοτήτων για τις αγορές, όπως επίσης ε, στο συντονισμό του ανεφοδιασμού. Ε, να πω ότι αυτό δεν συμβαίνει για την ώρα και ενδεχομένως ε, οι ζώνε δημοπράτηση και αναδιαμόρφωσή τους και αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί και να συζητηθεί για να έχουμε πιο ε, καλή διαμόρφωση των ζωνών αυτών δημοπράτηση. Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Θα δείτε περισσότερα στους τόμους που έχουμε δημοσιεύσει και που πρόκειται να δημοσιεύσουμε σύντομα. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, συνεργασία σας κατά τα τελευταία χρόνια από την αρχή του ενεργειακού πακέτου, δηλαδή από το 2010. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εξετάζεται όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Λάγκεν, που ήθελε να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθύντα. Συνολικά, ο οργανισμός έκανε πολύ καλή δουλειά. Ξέρουμε ότι αργά προχωρούμε, γιατί τα κράτη-μέλη μπορεί να μπλοκάρουν τις εξελίξεις ε, κάποια στιγμή. Οι διασυνδέσεις είναι δύσκολες, δύσκολο θέμα εδώ και καιρό. Στην αρχή της συζήτηση λέγαμε ότι οι διασυνδέσεις δεν είχαν γίνει δεκτής από, μεταξύ, και από μεγάλα και από μικρά κρατημέλη και ο ΆΣΕΡ έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει, να προωθεί τις διασυνδέσεις, να τις μεταφέρει και σε κάποια κράτη υπάρχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες αν δούμε τις ετήσιες εκθέσεις. Ε, πρόσεξα μια άλλη περίπτωση, την περίπτωση Ακβίντ, όπου ο γαλλικός οργανισμός δικτύων αναφερόμενοι στο Brexit που δεν το πιστεύω ότι και σίγουρο εγώ και στο βαθμό που νομικό και οικονομικό πλαίσιο δεν έχει ρυθμιστεί λέει ότι δεν μπορεί να λάβει απόφαση προτού δοθούν απαντήσεις όλα αυτά. Αυτό είναι θέμα κυρίως μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας και είδα ότι υπάρχουν πολλά θέματα εκεί. Βέβαια, το πρόγραμμα ωφελεί κυρίως στους Βρετανούς και αυτό είναι πολύ εντάξει γιατί θέλουμε να δράσουμε διασυνοριακά ακόμα και όταν ε, γίνονται διαπραγματεύσεις με την Βρετανία θέλουμε να ανοίξει αυτή η μεγάλη αγορά αλλά αυτές οι δομές λήψης αποφάσεων Αν ήταν στι εθνικές αρχές θα υπήρχαν περισσότερες καθυστερήσει. Ρωτώ λοιπόν εσάς. Πρώτον, υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές όπου δεν μπόρεσε να επηρεάσει ο Άσερ τι εθνικές διοικησει Και δεύτερον, στην περίπτωση Ακβίντ θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι δικαιολογημένο αυτό που λένε οι Γάλλοι η δήλωση δηλαδή του ρυθμιστικού φορέα ενέργεια είναι σωστή ή όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτροσον, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Ποτόσνικ για την εξαιρετική παρουσίαση και το καταπληκτικό έργο του οργανισμού υπό την ηγεσία σας. Πολύ το εκτιμούμε αυτό. Ε, αναφέρατε και κάποια νούμερα. Θα ήθελα να τα δούμε λίγο καλύτερα. Κατάλαβα για τα διασυνοριακά θέματα ότι είπατε ότι μισή, μισό δυναμικό το διασυνοριακό αξιοποιήθηκε πέρσι. Αυτό μοιάζει και με το προηγούμενο έτος. Αν λοιπόν κατάλαβα καλά, δεν γίνεται πρόοδος εις ό,τι αφορά τις διασυνοριακές ανταλλαγές. Συμφωνείτε? Τι άλλο μπορείτε να πείτε σχετικά με αυτό. Επίσης, η διαφάνειά σας ε, για τα επιδόματα, τα πιθανά επιδόματα ε, για, ε, για την πρόθεση των διασυνοριακών ανταλλαγών. Κατάλαβα καλά ότι αν προσθέσουμε αυτά τα επιδόματα πάμε κοντά στα 10 δις ευρώ το χρόνο σε επιδόματα για όλους τους Ευρωπαίους αν τα δώσουμε όλα ας πούμε είναι σωστό αυτό και πάλι ευχαριστώ για το εξαιρετικό έργο του οργανισμού και για το δικό σας προσωπικά ευχαριστώ πολύ Κύριος Δαλούντε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά γιατί μας περιγράψατε όμως μια ε, θλιβερή κατάσταση γιατί δεν ε, ανοίγουν τα σύνορά τους οι χώρες και μένουν στις εθνικές πολιτικές. Αυτό είναι κακά νέα ε, για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους γιατί πολλά χρήματα έχουν δαπανηθεί για την για τα διασυνοριακά δίκτυα, αλλά δεν έχουν τελικά τον θετικό αντίκτυπο. Τα κλειστά σύνορα δημιουργούν και προβλήματα προμήθειας. Ε, η μεγάλη κρίση μας δείχνει κιόλας τι μπορεί να συμβεί. Ίσως δεν σταματήσουν και οι διαπραγματεύσεις για τους νέους κανόνες. Ξέρουμε ότι ορισμένες χώρες ε, ε, θέλουν να συνεχίσει η κατάσταση όσο έχει, ενώ εμείς ως πράσινοι θέλουμε να μπουν σε νέα τροχιά. Θέλουμε ένα, μια υπηρεσία άσερε που θα είναι ισχυρή και ανεξάρτητη, ε, με έναν απολύτως αμερόληπτο διευθυντή που θα μπορεί σωστά να αξιολογήσει την κατάσταση. Ευελπιστούμε ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης θα καταφέρει να διαπραγματευτεί σωστά το θέμα ε, από πλευρά Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριο Σκόχλητς. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω ε, στο θέμα που είχαμε συζητήσει την τελευταία φορά με τον κύριο Ποτότσνικ. Όχι στη Βιέννη, αλλά στην Επιτροπή μας. Σε αυτήν λοιπόν την τελευταία συνεδρίαση είπαμε ότι όσον αφορά την ροή ηλεκτρικής ενέργειας πέραν των συνόρων υπάρχουν ε, χώρες, συγκεκριμένα η Πολωνία, που προσπαθούν να εμποδίσουν ακριβώς αυτήν την ροή εκτός των συνόρων. Ε, στην ε, Σιλεσία αλλά και σε άλλα σημεία της τσεχικής δημοκρατίας. Ε, η διασύνδεση είναι καλή αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε πέραν των συνόρων προς την Πολωνία. Επίσης στον χρωματιστό σας πίνακα με γκρίζο αναφέρεστε στις χώρες της Βαλκανικής αλλά δεν, δεν ξέρουμε εάν ε, ε, αναφέρεστε στην Βοσνία Ριζεγοβίνη ή στην Μακεδονία ή καλύτερα να πω στη Βόρεια Μακεδονία λέει ο μιλητής δεν ξέρω, έχετε διορθώσει λίγο την κατάσταση. Μας είπατε ότι οι χώρες αυτές υπερασπίζονται τα σύνορά τους και εμποδίζουν την ροή ενέργειας, το πέρασμα της ενέργειας, ε, πράγμα που έχει προκαλέσει προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Μπορεί να μας πει ο, ο, ο, ο μιλητής εάν θα βελτιωθεί το θέμα όσον αφορά τους αγωγούς και επίσης στο γράφημα για τα ποσοστά της 100 ε, εδώ έχουμε την, ε, την τιμή ε, συνολικά και με συμπεριλαμβανομένων και φόρων και ειδικών ποσοστών. Μήπως θα μπορούσε να μας δώσει κάποια στοιχεία αναχώρα. Πολλές ερωτήσεις λέει ο Πρόεδρος κύριε Διευθυντά. Μπορείτε να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που μου δίνουν την δυνατότητα να εμβαθύνω σε κάποια από τα σημεία. Ο κύριος Λάγκεν, αλλά και ο κύριος Πέτερσεν και άλλοι, έκαναν κάποια σχόλια. Είναι γεγονός ότι η προσόραση δεν χρησιμοποιεί χρησιμοποιούμε τους διασυνδετές, interconnectors με το πλήρες δυναμικό τους, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα ε, στις ε, διασυνοριακές ροές και τις εσωτερικές ροές. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση για την ηλεκτρική πραγματικότητα δεν απεικονίζεται σωστά. Είναι περισσότερο, απεικονίζεται περισσότερο στην ουσία η πολιτική βούληση. Υπάρχουν, τη Σουηδία, ε, ε, υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που δημιουργούν ε, που τα πράγματα πάνε καλά υπάρχουν και άλλες ζώνες ας πούμε εντός ε, των ε, ιδίων των χωρών όπου η κατάσταση δεν αντιπροσωπεύει την ηλεκτρική κατάσταση εκεί πρέπει να περιοριστούν οι ποσότητες που είναι διαθέσιμες στα σύνορα. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ επανέρχομαι στην άλλη του κ. Κόβετσεκ. Αυτό εξηγεί γιατί κάποια σύνορα ας πούμε, τα σύνορα μεταξύ της Γερμανίας, Πολωνίας, αλλά και της Γερμανίας με την Πολωνία και, της, ε, ε, και την Τσεχία έχουν ε, ικανότητα σχεδόν μηδενική, γιατί υπάρχει ικανότητα, αλλά πηγαίνουν στα λεγόμενα loop flows, που ε, έχουν ε, την ε, τάση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα λόγω τεχνικών προβλημάτων να σταματούν στα σύνορα και να διαχέονται στο εσωτερικό της χώρας. Γι' αυτό προτείναμε διάφορους τρόπους για να λύσουμε το θέμα αυτό. Πρώτον, μια καλύτερη δομή. Δεύτερον, ε, ε, σηματοδότηση αυτών που δημιουργούν, προκαλούν το πρόβλημα και επανεξέταση έτσι ώστε να δούμε τα ωφέλη και ε, τις ε, δυσχέρειες. Αυτό το είχαμε προτείνει ήδη τον Νοέμβριο του 2016 και αυτό ακριβώς κάνει και η Κομισιόν με την πρόταση διόρθωσης του Νοεμβρίου του 2016. Αυτό ακριβώς, αυτά είναι, αυτές είναι οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζει και ε, ο οργανισμός όταν, ε, αλλά τελικά δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε διότι οι δύο ρυθμιστικές αρχές δεν ε, συμφώνησαν ο Γάλλος ρυθμιστής, η Γαλλική ρυθμιστική αρχή και η ε, ε, Αγγλική ε, ρυθμιστική αρχή δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν το Άκεντ και μετά αυτό το θέμα ήρθε σε μας. Και μελετήσαμε πριν από ένα μήνα το θέμα αυτό και όπως είπατε υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο σύνορο αυτό και η αξιολόγησή μας, η εκτίμησή μας είναι ότι αυτός ε, ο Interconnector αλλά και άλλοι που έχουν αναπτυχθεί στα ίδια σύνορα ε, οπωσδήποτε θα είναι πολύτιμος αλλά θα είναι και ε, σωστός όσον αφορά την εξέλιξη του καθεστώτος των ρυθμιστικών αρχών αυτή τη στιγμή η ρυθμιστική αρχή της Γαλλίας δεν δίνει τέτοια δυνατότητα, αλλά αυτό είναι πρόβλημα γαλλικό και όχι πρόβλημα ευρωπαϊκής προσέγγισης. Κύριε Πέτερσεν, εδώ έχουμε κάποιες ε, εκτιμήσεις. Εάν δείτε υπάρχουν και κάποιες στήλες ε, ε, οι οποίες ε, δεν είναι το ίδιο πυκνές παντού, γιατί υπάρχει και ένα ε, σχετικό ποσοστό αβεβαιότητας. Η, ε, εμείς έχουμε ήδη περίπου πάνω από 15 δις όφελος, κέρδος. Τα στοιχεία μας είναι αρκετά αρκετά σωστά ε, και θεωρούμε ότι ε, με τον τρόπο αυτό ε, μπορούμε να προχωρήσουμε καλά. Φυσικά υπάρχουν ακόμα περιθώρια κέρδους. Κύριε Νταλούντε, σας είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη της, του οργανισμού μας. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να κλείσουν τα σύνορα. Αυτό είναι παράνομο βέβαια, αλλά δεν συμβαίνει και πολύ συχνά. Νομίζω άλλωστε ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε κάτι περισσότερο σε κάποιες ε, ε, περιοχές ναι, συμφωνώ με αυτό, αλλά από την άλλη μεριά ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ζήσουμε και με αυτά που έχουμε. Ο κύριος Κόβιτσακ επίση έκανε μια ερώτηση για τις βαλκανικές χώρες αλλά αυτές είναι εκτός της εντολής μας. Κάποια από τα στοιχεία τα οποία θα δείτε στο κείμενο καλύπτουν και αυτές τις χώρες, παρότι όμως ε, αυτές οι χώρες δεν συμμετέχουν ε, στην αγορά. Γίνεται μια προσπάθεια δημοπράτησης ε, της ικανότητας, αλλά δεν εφαρμόζουν το market coupling στον ηλεκτρισμό είναι γεγονός ότι πρέπει και αυτό το κομμάτι της Ευρώπης να οδηγηθεί προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν, είναι κλειστά τα σύνορα, ωστόσο δεν είναι ε, σε κατάσταση που να χρησιμοποιούνται όλοι οι πόροι με αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Νταμάτο, κοιτάξτε, όσον αφορά τους δασμού, τους φόρους, ε, μία σύνοψη για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο με τα διάφορα συστατικά των τιμών. Επίσης έχουμε και πληροφορίες αναχώρα λεπτομερή στον ε, τόμο που έχουμε εκδώσει. Εδώ βλέπετε στην αρχή τον ε, ΦΠΑ και μετά φόρους 23% για τον ηλεκτρισμό και περίπου το ίδιο ποσοστό για το φυσικό αέριο. Περίπου ένα πέμπτο έως ένα τέταρτο αφορούν φόρους. Ε, κύριε Λάγκε, σύντομα. Σύντομα, μια ακόμη ερώτηση για το ΑΚΒΙΤ. Είπατε ότι αυτή είναι μια απόφαση που μπλοκάρεται από τους Γάλλους. Τι θα γίνει, θα γίνει αγωγή κατά της Γαλλίας, παρέμβαση της Κομισιόν, ε, μεγαλύτερη παρέμβατική δυνατότητα από εσά. Τι λύση θα μπορούσε να βρεθεί για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Συγγνώμη, αλλά ίσως ε, ε, ε, δεν τα είπα εγώ καλά. Δεν λέω ότι μπλοκάρετε. Εμείς πήραμε την απόφαση και είπαμε ότι με τη δική μας ερμηνεία των διατάξεων, επειδή ο 437 του 2013 προβλέπει να παίρνει κανείς υποστήριξη και έγκριση. Αυτό λέει η Γαλλία. Και υπάρχει και νομολογία σε μας. Εδώ μπορεί να ισχύσει η εθνική νομοθεσία αν είναι σαφές ότι αντιβαίνει. Ε, ε, μπορεί να αλλάξει η εθνική νομοθεσία αν αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αν αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τότε Μπορεί ε, ε, να εξεταστεί πάλι το αίτημα για ε, απαλλαγή, για εξαίρεση. Θα πρέπει να δούμε αν συνάδει η γαλλική νομοθεσία με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά και συγχαρητήρια για τη σκληρή δουλειά σας. Ευχαριστούμε για την αφοσίωσή σας. Το τρίτο ενεργειακό πακέτο άρχισε με ε, και όλα τώρα είναι στα δικά σας χέρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, προχωρούμε και πάμε στο επόμενο σημείο που είναι το 19. Ε, ε, εκθέσεις για συνεχιζόμενες δια, διοργανικές διαπραγματεύσεις εσωτερική αγορά ενέργειας, Κοινή κανόνες για τους την εσωτερική αγορά ενέργειας. Στο δεύτερο ε, τριμερή διάλογο ήμουν εγώ, μπορώ να σας ενημερώσω σύντομα. Ο δεύτερος τριμερής, εκεί συζητήθηκαν κάποιες αρχές σχετικά με τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, άρθρο 3, επελεγμένα θέματα για τις αγορές την επόμενη μέρα και μέσα στη μέρα, άρθρα 6 και 7. Η επίδραση άρθρο 8 στις βράχη και μακροπρόθεσμες αγορές και προϊόντα. Ελάχιστο μέγεθος εμπορευομένων ε, προϊόντων. Το δεύτερο κομμάτι του τριμερούς διαλόγου ήταν αφιερωμένο στη, στα άρθρα 32 με 43, περιφερειακή συνεργασία. Η, τα θεσμικά όργανα έκαναν μια γενική συζήτηση σχετικά με τα βασικά πολιτικά θέματα που αφορούσαν τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού και τους ε, περιφερειακούς συντονιστές ασφαλείας. Αυτό το λέει το Συμβούλιο και αποφάσισαν να δώσουν εντολή για περαιτέρω εργασίες σε τεχνικό επίπεδο. Τώρα, ο δεύτερος τριμερής ε, διάλογος για την οδηγία διάφορες διατάξεις σχετικές με την ενίσχυση και την προστασία των καταναλωτών, δηλαδή ε, ποιες ε, συμφωνίες τιμών, ε, το switching, η αλλαγή ε, μέσα σύγκρισης, τιμολόγηση. Κάποιες συμβιβαστικές λύσεις πάνω σε αυτά τα θέματα έχουν επιτευχθεί, κάποια θέματα έχουν, επίμαχα θέματα έχουν λυθεί, αλλά παραμένουν ανοιχτά ακόμα. Οι διαπραγματευτές επίσης ενέκριναν προσωρινές συμφωνίες ε, που επετέφθησαν σε τεχνικό επίπεδο πριν από τον τριμερή διάλογο. Και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συζητηθούν ακόμη περισσότερο τα πράγματα σε τεχνικό επίπεδο. Και τα δύο θέματα, οδηγία και κανονισμό, θα συζητηθούν στον επόμενο τριμερή διάλογο στις 18 Οκτωβρίου του 18, σε 10 μέρες δηλαδή. Σημείο 21 ε, τιμότητα ανάληψη κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Φλάβιος Ζανονάτο είναι ο εισηγητής. Τι γίνεται λοιπόν στις δικές σας τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχαμε πολλές διμερείς ε, συμφωνίες ε, με την προεδρεύουσα χώρα της, ε, του Συμβουλίου αλλά και με την Κομισιόν πριν φτάσουμε στον πρώτο τριμερό, τρι, τριμερή διάλογο. Το κλίμα ήταν καλό. Έλαβε χώρα την 15η Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν βεβαίως αποστάσεις θέσεων, αλλά υπάρχουν τρία στοιχεία επί των οποίων συμφωνούμε το ε, μοντέλο template, ε, η κατεξουσιοδότηση πράξης, ε, καθώς επίσης και η εισαγωγή κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά την αμοιβαία αρρωγή, καθώς επίσης και τον έλεγχο εξάντε της Κομισιόν επί των ε, εθνικών ε, μεθοδολογιών. Ε, ο έλεγχος είναι ο μόνος τρόπος, ο έλεγχος των εγκαταστάσεων είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε καλά συγκρίσιμα στοιχεία. Το Συμβούλιο θέλει να αφήσει τα κράτη-μέλη ελεύθερα ε, να καθορίσουν ε, ε, σχέδια και εγκαταστάσεις. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα στα οποία έχει εξουσίαση η Κομισιόν, τα σημεία 13 και 19, για το μοντέλο αυτό δεν θα υπάρξει ανάγκη τροποποιήσεων γιατί ρυθμίστηκαν κατά θέματα στον πρώτο τριμερή διάλογο. Ε, ε, βάση του εγγράφου καθορίζονται ε, σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την συνεργασία, ωστόσο δεν καθορίζονται τρόποι εφαρμογής, κυρίως όσον αφορά την καλή αποζημίωση. Ε, υπάρχει ζούγκλα πραγματική όσον αφορά και πληθώρα εν πάση περιπτώσει δυνατοτήτων και συστημάτων και μεθοδολογιών αποζημίωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε ε, οπωσδήποτε να υπάρξει κάποια καθοδήγηση. Το ε, Συμβούλιο όμως ε, είναι διστακτικό, μιλάει για υπερβολική γραφειοκρατία. Το σημείο στο σημείο 3 ε, οι θέσεις ε, είναι ακόμα πολύ απομακρυσμένες το, το Συμβούλιο δεν προτίθεται ε, να ε, καλύψει την δυνατότητα προληπτικής παρέμβασης της Κομισιόν. Από τη δικιά μου μας πλευρά λέμε ότι ο Ευρωπαίος ε, νομοθέτης πρέπει να έχει κάποια εργαλεία στην διάθεσή του εάν θέλει να είναι σίγουρος για την καλή λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής συγγνώμη αγοράς σε αγαστή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και βεβαίως και σε σχέση με τις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια. Θα μπορούσαμε να ε, δούμε κάποιες δυνατότητες οι οποίες δεν αμφισβητούν την δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίζει, αλλά ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν οι μεθοδολογίες που ακολουθούν ε, τα, οι διάφορες εγκαταστάσεις στην γενικότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των ε, στοιχείων τα οποία ε, περιλαμβάνονται στον κανονισμό ε, οι διατάξεις για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση και η εμπλοκή των όλων των εμπλεκομένων φορέων στην, στον καθορισμό ορθών μεθοδολογιών είναι πράγματα πολύ σημαντικά. Επίσης, ε, οι τεχνικοί σύμβουλοι εργάζονται ήδη ε, αυτή τη στιγμή, ενώ στο Στρασβούργο στις 23 Οκτωβρίου προβλέπεται επόμενη συνεδρίαση. Ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να κλείσουμε σωστά τον ε, επόμενο τριμερή διάλογο και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λάγκεν. Ένα γενικό σχόλιο. Um, ο κύριος Πέτερσεν Μπορείτε να μας παρουσιάσετε Ναι υπάρχει Υπάρχουν διαπραγματεύσεις ε, τριμερείς Κάνουμε πρόοδο Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε Έχουμε πολλές συζητήσει να κάνουμε σε τεχνικό επίπεδο και ελπίζω να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο μέχρι το δεύτερο τριμερή διάλογο που θα γίνει στις 23 Οκτωβρίου. Ε, ακούσαμε και την παρουσίαση του κυρίου Ποτότσνικ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που ακούσαμε από τον κύριο Ποτότσνικ ε, για να μπορέσουμε να ε, βοηθήσουμε αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που χρειάζεται για να υπάρχει αυτή η ρυθμιστική εποπτεία με την οποία έχει επιφορτιστεί ο Άσερ. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας και πρέπει εδώ στο Κοινοβούλιο να συνεργαστούμε ε, και με το Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα όμως ε, που είναι τεχνικού επίπεδου και ελπίζω να μπορέσουμε να σημειώσουμε ε, πρόοδο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου που είναι ο επόμενος τριμερής διάλογος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεν. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το κανονισμό. Δεν, δεν ήθελα να πω για το να σε... Μια γενική παρατήρηση ήθελα να κάνω μετά τους πολυμερείς ε, διαλόγους στην Οικονομική και τη Βιομηχανική Επιτροπή. Είμαι 24 χρόνια μέλος του Κοινοβουλίου και διαπιστώνω ότι ε, μειώνεται η δύναμη των ομάδων γιατί αποδυναμώνονται και οι ε, βουλευτές. Δεν το λέω προς, τη, τον εισηγητή, αλλά είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Ε, πρώτη ε, αιτίαση. Όταν γίνονται διαπραγματεύσεις Κοινοβουλίου-Συμβουλίου θα ήταν αρκετό να ρυθμίζαμε και να λύναμε τα πολιτικά ζητήματα με διαφορετικά μέτρα και από τη διοίκηση. εντωμεταξύ έχει αυτό εκφυλιστεί σε ε, μία σχολαστική δραστηριότητα και αναλωνόμαστε σε προβλήματα που θα μπορούσαν να λυθούν σε τεχνικό επίπεδο και δεν λύνουμε τα πολιτικά. Γιατί σημαίνει αυτό. Είναι πολύ λεπτομερής ο ε, σχεδιασμός. Έχουμε κρίσιμα ζητήματα, ένα, δύο, τρία μάξιμουμ μπορεί να λυθούν. Έχουν προβλεφθεί τέσσερις ε, τριμερείς διάλογοι, τέσσερις σχεδόν πέντε τεχνικοί ε, ε, διάλογοι και πέντε προπαρασκευαστικές συναντήσεις για τους, για τις, τις, τους τεχνικούς ε, τριμερείς διαλόγους. Ε, τελευταία συνεδρίαση έγινε από τους Σκιώδης 25 Σεπτεμβρίου. Ακόμα προβλέπονται 14 συνεδριάσεις όλων αυτών ανεξάρτητα από την πορεία της συζήτησης. Αυτό οφείλεται σε, πολλού πολλούς λόγους. Πρώτον, στις ε, γραμματείες είναι ένας συνεργάτης υπεύθυνο για ένα φάκελο και πρέπει να αποδείξει τη δουλειά του, ένας αναφάκελο. Νομίζω ότι έτσι ε, επιβαρύνονται οι βουλευτές, ε, πέφτουν σε γραφειοκρατία και δεν μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους καθήκοντα. Αυτό δεν παρατηρείται μόνο εν προκειμένου, αλλά και Επίσης το Συμβούλιο όλο και λιγότερο ε, συζητεί με εμπειρογνώμονες που είναι και σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Αν το, αν το Συμβούλιο δεν ε, προσωπείται από υπουργούς, από πολιτικό προσωπικό, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Ε, δεν ε, Υπάρχουν ειδικοί εμπειρογνώμονε, όχι όμως εξουσιοδοτημένοι να λάβουν πολιτικές αποφάσεις και έτσι δεν προχωράει το πράγμα. Όλο λένε θα ρωτήσουμε το Συμβούλιο. Δεν μπορεί να γίνονται έτσι διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο. Τρίτον, έχουμε συνηθίσει να μην παίρνουμε πρώτα τη θέση μας στο Κοινοβούλιο και μετά να διαπραγματευόμαστε, αλλά να το κάνουμε αυτό πάνω στη βάση των ψηφοφοριών των επιτροπών. Και το λέω αυτό ως εκπρόσωπος της μεγαλύτερης ομάδας. Δεν επιτρέπεται οι αποφάσεις να λαμβάνονται από 8 σκιώδεις ε, ενώ ορισμένοι υποεκπροσωπούνται. Ε, και έτσι υπάρχει ε, μεγάλη πίεση για συμβιβασμό πριν γίνει ψηφοφορία στις επιτροπές καν. Αυτό δεν έχει να κάνει με τους ε, εισηγητές μας κάθε φορά. Είναι μια γενικότερη ε, έλλειψη, μια δυναμία που πρέπει να την απαλείψουμε. Και η Κομισιόν σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων μόνο γνωμοδοτεί. Βεβαίω έχει το δικαίωμα να αποσύρει τις προτάσεις της και να υποβάλει καινούριε, αλλά δεν λαμβάνει αποφάσεις. Και κάποιοι ε, υπάλληλοι της Κομισιόν θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, οφείλουν να ακολουθούν την Κομισιόν. Αυτά είναι γενικότερα προβλήματα που ήθελα να τα αναφέρω σήμερα. Εσείς υπήρξατε και πρόεδρος του Κοινοβουλίου σε εποχές που δεν ήταν τόσο δυσάρεστες. Ε, σε εποχές που δεν ήταν τόσο Ελπίζω να ε, μ' ακούσετε προσεκτικά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις σας γιατί είναι γενικές και πολύ σοβαρές Πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα μπροστά μας. Η Επιτροπή μας ε, συμμετέχει σε 17 διαπραγματεύσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για τη γραμματεία, για τους συμβούλους των πολιτικών ομάδων να τα χειριστούν όλα παράλληλα. Εν πάση περιπτώσει, α, θα λάβουμε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις σας. Εγώ δεν βλέπω το πρόβλημα ως τόσο σοβαρό ε, όσο εσείς, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το σκεφτώ. Και πράγματι, και μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε. Κάποια σημαντικά στοιχεία που σας απασχολούν τα λάβουμε υπόψη μας. Μήπως, ε, Μόρτεν, θες να πεις τίποτα? Όχι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστέ οι παρατηρήσει σου και δεν έχω την εμπειρία του κυρίου Λάγκεν για να μπορέσω να κρίνω ή να καθαρίσω πώς ήταν η κατάσταση πιο πριν, αλλά μπορώ να διαβεβαιώσω όλους σας ότι θα προσπαθήσουμε να δράσουμε ταχύτατα ε, λόγω των ημερομηνιών. Αυτή είναι η φιλοδοξία, να το ολοκληρώσουμε και τα χρονοδιαγράμματα, αν κατάλαβα, είναι δύσκολα. Έχουμε καθυστερήσει, πρέπει και να συνεργαστούμε και με το Συμβούλιο και δεδομένων των εντολών είναι δύσκολα τα πράγματα. Κανείς δεν θέλει να παραταθούν οι διαπραγματεύσεις αυτές, αντιθέτως. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Οπότε ας προσπαθήσουμε να κινηθούμε με ε, βάση αυτές μας τις φιλοδοξίες. Ναι, θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα και για κάθε διάλογο. Συνάδελφε, έχετε το λόγο. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια γενική συζήτηση από τους συντονιστές. Θυμάμαι την προ προηγούμενη θητεία Υπήρχαν δύο σημαντικά θέματα. Στη μία περίπτωση ο Ολλανδός ε, Υπουργός Οικονομικών Ντάισελ Μπλουμ στη συνεδρίαση ε, συμφώνησε σε πολιτική συμφωνία κατα, ε, ε, ε παρακάμπτοντας τους ε, υπαλλήλους. Ο δεύτερον, ο Γάλλος Υπουργός Περιβάλλοντος Πολό είχε πει ότι θα επιβάλλω τα θέματα αυτά στη χώρα μου. Αν δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό, αλλά μόνο οι υπάλληλοι, τότε διαιωνίζονται οι διαπραγματεύσεις. Το Κοινοβούλιο σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να συζητά ισότιμα με το Συμβούλιο και να μην χάνεται σε τεχνικές λεπτομέρειες και αυτό πρέπει να το σημειώσει και να συμμορφωθεί και η Γραμματεία. Εντάξει, ναι, συμφωνούμε μαζί σας. Ενδεχομένως τα προβλήματα που βλέπετε εσείς ε, ως πολύ σοβαρά, εμείς να μην τα βλέπουμε ως τέτοια. Θα το λάβουμε βέβαια υπόψη είναι αυτά που μας είπατε. Ε, πολλές συζητήσεις γίνονται σε τεχνικό επίπεδο. Πάρα πολλά ζητήματα έχουμε σε τεχνικό επίπεδο. Μόρτεν είπε ε, στην περίπτωση του πρώτου τριμερούς ε, ε, διαλόγου κάποια ζητήματα που αφορούσαν το Acer τελικά πρέπει να επιληθούν σε τεχνικό επίπεδο. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη κάποιες από τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγα λεπτά θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας στην κοινή με την Επιτροπή Μεταφορών. Περιμένουμε τους συναδέλφους μας.